Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας καλωσορίσω στη σημερινή συνεδρίαση. Σας καλησπερίζω. Σήμερα έχουμε πολλά μεγάλα γεγονότα. Θα ήσασταν κάποιοι στην συνδιάσκεψη των Προέδρων με τον Πρόεδρο Βαρόζο και με τον Πρόεδρο Φαν Ρομπάι. Επίσης, παρόν ήταν και ο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Μάριο Ντράγκη. Σήμερα εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα ασχοληθούμε με πολύ βαθιά ζητήματα και σοβαρά της δαπάνης κονδυλίων. Δεν είναι ασήμαντο αυτό που κάνουμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν όλοι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, επιθυμίες για αλλαγή στην εμερήσια διάταξη. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Οπο... Α, κι όμως ο κύριος Ρούμπιχ θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, πρόεδρε. Ήθελα να πω μόνο ότι συνήθως οι, συνδυα... οι συνεδριάσεις μας πάνε μέχρι τις 6.30 και ίσως ε, πολλοί, από την, ε, πολλοί συνάδελφοι να έχουν ε, κάποιες υποχρεώσεις από τις 6.30 και μετά. Και εγώ δυστυχώς 6.30 ώρα έχω ένα άλλο ραντεβού, μια άλλη υποχρέωση. Οπότε αν θέλετε να είσαστε λίγο αυστηρός με το χρονοδιάγραμμα για να προχωρήσουμε όσο γίνεται μέχρι εκείνη την ώρα. Ωραία. Αυτό βεβαίως ισχύει για όλους. Επομένω, ε, θα μπορούσαμε ίσω και τον ε, χρόνο ομιλία να τον ε, μειώσουμε στο μισό. Σα ευχαριστώ που μου το είπατε κύριε Ρούμπι. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται και στο ίντερνετ. Επίσης να πω ότι η Επιτροπή μας προσεκλήθη να χρησιμοποιήσει ένα νέο application και το είχαμε ξαναπεί ε, και βεβαίως ε, ευχαριστούμε και τη Γενική Διεύθυνση ITEC που μας ε, προσκόμισε το νέο application για το e-meeting. Λοιπόν, πάμε στην έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης των 10 Ιανουαρίου, 21-27 Ιανουαρίου και 24 Ιανουαρίου. Σας έχουν αποσταλεί με email, δεν βλέπω να υπάρχουν αιτήσει για κάποια αλλαγή, εγκρίνονται λοιπόν και τα πρακτικά. Πάμε στην απαλλαγή 2011 Γενικός Προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισηγήτρια, η Εύα Ορτής Βιλέγια, είναι εδώ και θα δούμε το σχέδιο της νομοδότησης. Παρακαλώ, η εισηγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν συνοψίσω τις δασικά σημεία, τη εκθέσεω όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2011. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του συντρόφου για την υποστήριξή του και τι προτάσει του όσον αφορά το κείμενο, κυρίω οι συγητέ οι όσοι συγητέ. Και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε από τη στιγμή που θα έχουμε στα χέρια μα τι διάφορε τροπολογίε που αφορούν το κείμενο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης για τις απαντήσεις και που μας έδωσε ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Μπελέν, που πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα μας απαντούσε και ήρθε τον περασμένο μήνα στην Επιτροπή μας για να απαντήσει στις ερωτήσει που ε, ε, του θέταμε, ε, καθώς ευχαριστώ και τις διάφορες γενικές διευθύνσεις, οι οποίες μας έδωσαν διάφορες απαντήσεις και μας επέτρεψαν να ετοιμάσουμε ακριβέστερη έκθεση θα ήθελα να αναφέρω επίσης και τη συνεδρίαση που έλαβε χώρα με, τη, με την ε, συμμετοχή του εσωτερικού διατάκτη ε, που μας οδήγησε μια αποκαρποφόρα συνεργασία και ευχαριστώ και τη γραμματεία της Επιτροπής μας καθώς και τους διοικητικούς που είναι υπεύθυνοι για το θέμα, καθώς και την ομάδα που παρακολούθησε όλες τις εργασίες, όπως είπα, στις 23 Ιανουαρίου, με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζητήσαμε και στόχος μου ήταν να φροντίσουμε ούσο ώστε τα, τα χρήματα, τα δημόσια του φορολογούμενου να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, ε, θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια έκθεση όσον αφορά την απαλλαγή που θα ήταν επικοδομητική, που θα οδηγήσει σε συνένεση και έτσι σε αυτό το πνεύμα συνεργάστηκα με τους διάφορους που προανέφερα για να σας δώσω αυτό το έγγραφο που έχετε μπροστά σας. Αυτή η έκθεση δεν θα αποφύγει τις διάφορες κριτικές που είναι απαραίτητες, είναι αναγκαίες. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η καρδιά της δημοκρατίας στην Ευρώπη και εκπροσωπεί 500 εκατομμύρια πολίτες και θα πρέπει να δίνει παράδειγμα όσον αφορά τον λεπτομερή έλεγχο των δαπανών. Σε αυτή τη φάση μάλιστα τώρα όπου περνάμε μια σοβαρή οικονομική κρίση τη στιγμή όπου οι πολίτες της χώρας μας πρέπει ε, να επιδείξουν αποτελεσματικότητα στον αφορά των χρημάτων και ορθολογιστική προσέγγιση. Θα πρέπει εδώ να δείξουμε ότι τους υποστηρίζουμε όντας αποτελεσματικοί στην καθημερινή μας δουλειά. Η διαχείριση του προϋπολογισμού είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό συνεπιφέρει προσπάθεια για διαφάνεια και ευθύνη και αποτελεσματικότητα. Και γι' αυτό και το θέμα των δημοσίων προμηθειών και το πλαίσιο το σωστό θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου. Και γι' αυτό στην έκθεση που υποβάλλω τονίζω ακριβώς αυτά τα θέματα των δημοσίων προμηθειών. Εξάλλου θα μπορείτε να παρατηρήσετε ίσως στην έκθεση αυτή ότι αναφερόμαστε στην ε, ευφυή εξοικονόμηση. Θέλουμε να κάνουμε οικονομίες, αλλά οι προσαρμογές αυτές δεν θα πρέπει να έχουν συνέπειες όσον αφορά τους πόρους που επηρεάζουν τις αστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε εξορθολογιστική χρήση των χρημάτων, αποτελεσματική χρήση των διαθεσίμων πόρων. Ένα άλλο θέμα επί το οποίο επιμένουμε και είναι κάτι που μας ανησυχεί είναι η ασφάλεια. Ε, κάποιοι συνάδελφοι έχουν προβλήματα με κλοπές στα γραφεία τους. Το 2011 το Προεδρείο υιοθέτησε τη νέα αρχή, τη νέα έννοια της γενικής ασφάλειας, καθορίζοντας διάφορες περιμέτρους ασφαλείας, γενικές, γενικές περιμέτρους ασφαλείας, που θα πρέπει να εγκριθούν από το Προεδρείο. Εδώ θέλουμε να τονίσουμε και το, την εσωτερική του χρέους των υπηρεσιών ασφαλείας. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια που επικρατεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άλλο σημείο αφορά τα, τα πορίσματα της ετήσιας ε, έκθεσης του εσωτερικού ελεγκτού όσον αφορά καλύτερο σχεδιασμό που απαιτείται. Η έλλειψη σχεδιασμού οδήγησε στο ότι κάποιες διευθύνσεις, κάποια τμήματα έπρεπε να περάσουν μέσα από έκτακτες διαδικασίες ε, για ε, δημοσίες προμήθειες. Τονίζεται εδώ επίσης ε, ε, τονίζονται οι διάφορες εξωτερικές συμβάσεις που έχουν συνάψει οι διάφορες γενικές διευθύνσεις. Αναφέρονται επίσης και τα προβλήματα τα δομικά ε, του ημικυκλίου, του, του, της έσωσης του Αυγούστου 2011 και ότι χρειάζεται να προγραμματιστούν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν για να αποκατασταθεί το ημικύκλιο. Στην έκθεση επίσης λέμε ότι το 2011 γιορτάσαμε τελευταία φορά ε, το βραβείο, την απονομή βραβείου για τη δημοσιογραφία, κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής μας. διότι το κόστος αυξήθηκε, οι δαπάνες αυξήθηκαν και χρειάζεται περικοπή των δαπάνων. Αναφέρουμε επίσης και όσα αφορούν και το Γραφείο Ταξιδίων, 31 Δεκεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, εκπνέει το συμβόλαιο, η σύμβαση και ζητώ στην έκθεση αυτή όχι μόνο να κάνουμε οικονομικό έλεγχο, αλλά έλεγχο της δομής και της επίδοσης του ταξιδιωτικού γραφείου. Αυτές είναι οι βασικές γραμμές που ακολουθεί η έκθεσή μου όσον αφορά την απαλλαγή για το 2011 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για μία ακόμη φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για τη συνεργασία σας. Περιμένω τροπολογίες σας και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Πρώτα να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο Γκέρμπραντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή. Όχι μόνο για την έκθεση, αλλά για τον τρόπο επίσης με τον οποίο μπορέσαμε να συνεργαστήκαμε. Η συνεργασία ανάμεσα στο, σε αυτόν και στους εισηγητές. Παρ' αυτά, μια μικρή παρατήρηση να κάνω αν επιτρέπετε. Περνάμε μια δύσκολη περίοδο από δημοσιονομικής απόψης και πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί όσον αφορά τις δαπάνες, τις που κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Για, αυτό το λέμε για το 2013, αλλά αυτό πρέπει να ισχύει και το 2012, κάτι που κάνουμε τώρα ε, με τον έλεγχο. Θα πρέπει δηλαδή να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το μέλλον. Τώρα, κάποια στοιχεία. Παράγραφος 1 για τη διαφάνεια. Συμφωνώ. Υπάρχει όμως κάτι που λείπει. Ίσως δικαιολογημένα. Είχαμε το αίτημα να γίνει μια συζήτηση στην Ολομέλεια για την απαλλαγή με τον Πρόεδρο. Αυτό να γίνεται θυσίως δηλαδή. Αυτή, αυτός ο διάλογος για τη διαφάνεια είναι σημαντικό και θα πρέπει ο, όχι μόνο αντιπρόεδρε αλλά ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου να αναλάβει την ευθύνη του και να δει το θέμα που έχει να κάνει με τις απάντες. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω το εξή. Αν είναι δυνατό εξ ονόματι της Επιτροπής μας να συντάξετε μια ε, επιστολή για τη διάσκεψη των Πρόεδρων υπενθυμίζοντας το, το ψήφισμα το περσινό δηλαδή της οργάνωσης μιας ολομέ συζήτηση στην Ολομέλεια για το θέμα της απαλλαγής. Κάποια στοιχεία ακόμα να πω, να προσθέσω. Υπάρχουν κάποια πράγματα που λείπουν κατά μένα. Ε, εδώ και δύο χρόνια ζητήσαμε να υπάρχει ένας ηλεκτρονικός έλεγχος ε, για τα μέλη του Κοινοβουλίου. Δεν είναι δύσκολο. Υπάρχουν ήδη δυνατότητες και θεωρώ ότι είναι άδικο ότι όλοι, όλοι μπορούν να ε, περάσουν από κάποιους αυτόματους ε, ε, από την αυσόρδα αυτόματα, με αυτόματο τρόπο, αλλά όχι οι βουλευτές. Αυτό ίσως θα πρέπει να το δούμε και θα μπορούσαμε ίσως να το διευθετήσουμε. Κάτι άλλο. Η μείωση του όγκου του χάρτην όγκου. Ε, βλέπετε μια φύσα που ε, γίνεται μια ανακοίνωση για κάποια συνάντηση. Ε, εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζομαι πλέον χαρτιά εδώ και εκεί. Αλλά τι γίνεται, φτάνω εδώ πέρα και δεν βλέπω 20 εκατοστά ε, τα έγγραφα τα οποία είναι μπροστά μου. Θα πρέπει να το δούμε με, τις, ε, με τους αρμόδιους, ούτως ώστε να μην τυπώνονται άλλο τα έγγραφα αυτά να βρούμε ένα άλλο τρόπο. Ένα άλλο στοιχείο επιπλέον, το οποίο δεν το βλέπω στην έκθεση, στο σχέδιο μάλλον της έκθεσης, είναι αυτό που ονομάζω για, για την αποζημίωση που έχουμε για τα γραφεία μας. Δεν είναι επίκαιρο πλέον αυτό το θέμα. Εγώ θα καταθέσω τροπολογία πάνω σε αυτό το θέμα, σας το λέω τώρα εδώ για να μπορέσουμε. Για να, για να δικαιολογεί κανείς, ε, να μπορεί να δικαιολογήσει και να έχει αποδεικτικά στοιχεία ε, για κάθε δαπάνη. Επίσης, εγώ θα ήθελα να πω, είμαι, εντυπωσιάζομαι, δηλαδή μου προκαλεί έκπληξη το Προεδρείο καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα συνεχώς σε σχέση με αυτά τα οποία καταλήγουμε εμεί στην Ολομέλεια Φερρυπίνα. Μήπως θα πρέπει να ενισχυθεί εδώ, εδώ πέρα η, ορο, ε, ορολογία, τι ακριβώς χρησιμοποιούμε. Επίσης, κάτι άλλο που παρατήρησα τα τελευταία χρόνια για τα υποχρώσεις της, ε, σε σχέση με το πρωτόκολλο που έχουμε. Ε, υπάρχουν διαφοροποίησεις εδώ ανάλογα με τα μέλα του Προεδρείου. Πολλά μέλη δεν συμβάλλουν ε, σε εργασίες των αντιπροσωπιών και αυτό κοστίζει πολύ. Συχνά βλέπουμε κάποιες ε, αποστολές σε απομακρυσμένες, ε, απομακρυσμένους προορισμούς. Θα μπορούσε κανείς να έχει εναλλακτικές λύσεις και για να μην γίνονται όλες αυτές οι δαπάνες. Τώρα, κάτι τελευταίο. Η Επιτροπή Επιτροπού, ε, προπολογισμού τα 2012-2013 ζήτησε μια αξιολόγηση εξωτερική του προπολογισμού του δικού μας. Έχουμε πληροφορίες από τους δικούς μας τους υπαλλήλου και πραγματικά αυτό πολλές φορές ε, διαψώνει κανείς ότι ορισμένες δαπάνες δεν είναι και τόσο απαραίτητες. Ίσως να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι να, ούτως ώστε να έχουμε μια, ένα οργανισμό εξωτερικό ο οποίος θα μπορέσει να ελέγξει το προπολογισμό μας και να δει μήπως μια σειρά στοιχείων όσον αφορά το προπολογισμό μας είναι, είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να κοιτάξουμε και με τον τρόπο να μειώσουμε τις δαπάνες μας. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Σαν κλείνω εδώ με τις πρώτες μου παρατηρήσεις και ανυπομονώ να ακολουθήσω τη συνέχεια του έργου μας. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο μόνο για τα ερωτήματα που θέσατε. Με, σε συζητήσεις που είχα με τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου προβλέπεται μία ξεχωριστή συζήτηση στην Ολομέλεια για την ε, απαλλαγή για, τον, για το Κοινοβουλίο. Αποφασίστηκε αυτό και από το τελευταίο ψήφισμα. Ε, ζήτησαμε λοιπόν να μάθουμε τι γίνεται και μας επιβεβαίωσαν ότι προβλέπεται να γίνει μια τέτοια έξτρα επιπλέον επιμέρους συζήτηση για, για την απαλλαγή. Επόμενος, ο συνάδελφος Δε Γιούγκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και τον κύριο Γκερμπράντη να ευχαριστήσω φαίνεται να έχει προσέξει, να έχει ενημερωθεί για τις παρατηρήσεις μου, για τα σημειώσει τι δικέ μου, γιατί ε, τα έχω όλα αυτά, ο, λέξη προς λέξη από αυτά που, αυτά που είπε. Λοιπόν, ε, τον υποστηρίζω τον καλ... πλήρως. Υπάρχει επίσης κάποιο άλλο σημείο, το οποίο θέλω να θίξω. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα στους πολίτες, υπάρχουν τα θέματα των αποζημιώσεων εν γέννη, και για μας. Ξέρω ότι υπάρχουν αντιπροσωπείες που είναι υπεύθυνε. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω. Κάθε μήνα ε, γίνονται δαπάνες, ε, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια τροπολογία πολύ ε, δυνατή. Θα το κάνω εγώ αυτό, θα την καταθέσω. Διότι κανείς δεν μου εξήγησε. Και πραγματικά απευθύνθηκα σε πάρα πολλούς ε, για θέματα αποζημίωσης, για κάποιες αποζημίωσεις ε, λόγω αποστάσεως. Τι είναι ακριβώς αυτή εδώ αποζημίωση. Θεωρώ ότι σε θέματα ελέγχου του προπολογισμού, σε αυτό το θέμα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς ακριβώς δαπανούνται ορισμένα κονδύλια. Συμφωνώ πλήρως με την άποψη του κύριου Γκερμπράντη, του συναδέλφου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προσέχουμε ε, για το κοινό μας, για τους πολίτες. Θα πρέπει να δικαιολογούνται οι δαπάνες και έχει να κάνει αυτό με το κύριο μας και με την εικόνα μας. Όλες οι πληροφορίες δεν φτάνουν και η ενημέρωση δεν φτάνει μέχρι το, τον τελευταίο πολίτη. Πραγματικά. Να καταλάβουμε ότι το κείμενο είναι ελαφρύ κατά κάποια άποψη και δεν οδηγεί σε εξυγίανση που θα λέγαμε. Θα πρέπει να ενισχυθεί αυτό το κείμενο. Το ίδιο και για τον Ευρωπαϊκό ε, ε, για τον Νίκο για την ευρωπαϊκή ιστορία. Δεν θα πω τώρα σε λεπτομέρειες όμως. Συνολικά ε, είναι σαφέ ότι εγώ θα πρέπει να καταδέσω μια σειρά τροπολογιών. Παρόλο που συμφωνώ με αυτά που είπε ο εισηγητή σε γενικέ γραμμές ε, και συμφωνώ και είναι πολύ ε, ξεκάθαρες οι, οι θέσεις του, της θα πρέπει όμως να δούμε και άλλα θέματα που έχουμε να κάνουμε με εξοικονόμηση πόρων. Συμφωνώ με τι θέσει λοιπόν τη ηγετρία, αλλά για μια σειρά άλλων θεμάτων έχω ανακαταθέσει τροπολογίε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Ντεγιόγκ. Γκαρίγα, επόμενο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της, αλλά θα θέσω και ένα ερώτημα και έχω και μια παρατήρηση του σημείου 50. Αυτό αφορά την πολιτική για τα κίνητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τα δομικά προβλήματα που για δεύτερη διαδοχική φορά διαπιστώθηκαν, συνέβησαν προβλήματα στο ημικύκλιο χώρος που έχει ιδιαίτερο ρόλο για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Είχαμε πρόβλημα στο Στρασβούργο και έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα και για άλλη μια φορά στις Βρυξέλλες κάτι που επηρεάζει άμεσα ε, τη διεξαγωγή των ολομελιών μας. Βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να οργανώσουμε ολομέλειες στις ε, Βρυξέλλες και το κόστος για τις επισκευές είναι πολύ μεγαλύτερο από τις οικονομίες που κάνουμε εδώ και χρόνια όσον αφορά τους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια αυτό το θέμα να αντιμετωπιστεί με πιο αυστηρό τρόπο. Να αντιμετωπιστεί πιο αυστηρά η δίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν ζητάμε ε, απόδοση ευθυνών. Θέλουμε να δούμε γιατί σε 20 χρόνια τα δύο ημικύκλια είχαν προβλήματα δομικά, σημαντικά προβλήματα δομικά και κατασκευαστικά και ποιου μηχανισμούς έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτως ώστε τα χρήματα του φορολογουμένου να μην ε, πληρώνουν για ε, εσφαλμένες κατασκευές. Κατασκευές που σε λιγότερο από 20 χρόνια παρουσίασαν προβλήματα. Ε, νομίζω ότι έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα του φορολογουμένου και γι' αυτό θα ζητούσα από την εισηγήτριά μας να είναι πιο σκληρή στις συστάσεις που κάνει όσον αφορά τη συγκεκριμένη παράγραφο και κυρίως όταν ζητάει και άλλες πληροφορίε. Ε, Επόμενος, Γκάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την επιθυμία του κυρίου, μετά από την επιθυμία μόνο του κυρίου Ρούμπιχ, δεν θα πω όλα όσα ήθελα. Οι συνάδελφοι ήδη είπαν κάποια από τα σχόλιά μου. Εγώ εκπροσωπώ και τον ε, ε, ε, σκιώδη ηγητή, ο οποίο δεν μπόρεσε να έρθει από την ε, Ρουμανία, αλλά μου με ενημέρωσε ότι για, ε, το σχέδιο κειμένου της κυρία Ορτή δεν έχουμε, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, δεν θέλουμε να υποβάλουμε τροπολογίε. είναι καλή δουλειά που έκανε, είναι καλή η έκθεσή τη. Θα ήθελα μονάχα να πω δύο πράγματα για όλου όσου μίλησαν. Ε, έχουμε κάνει ε, πολλές συζητήσεις ε, επί του θέματος. Εγώ από τότε που είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής συνέχεια ακούω συζητήσεις που γίνονται σε τότε την Επιτροπή αλλά που τελικά εκτός αυτής δεν, δεν, έχει, δεν έχουν κανένα ρόλο να παίξουν. Η τηλεόραση, α πούμε, του Κοινοβουλίου, που έχει τύχει μεγάλης κριτικής και οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, ουσιαστικά πολλοί συνάδελφοι λένε ότι δεν παρακολουθούν την τηλεόραση του Κοινοβουλίου. Αν όμως ε, το δούμε πιο προσεκτικά, θα δείτε ότι πάνω από 20 κανάλια, πάνω από 20 χώρες ε, της Ευρώπης χρησιμοποιούν εικόνες από την τηλεόραση του Κοινοβουλίου. Δηλαδή φτάνει η κοινοβουλευτική τηλεόραση στις οθόνες των των πολιτών. Αν θεωρούμε ότι δεν είναι σημαντική η τηλεόραση του Κοινοβουλίου, τότε να αναρωτηθούμε αν όντω χρειάζεται και αν δεν χρειάζεται να δράσουμε αναλόγω. Μετά, το General Allowance. Ε, και για τούτο το θέμα έχουμε διαφορετικές ε, παραδόσεις ε, στην Ευρώπη. Ξέρω ότι υπάρχει μια χώρα και δεν είναι οι κάτω τις οποίες οι βουλευτές της πάντα λένε ότι αρνούμαστε να κάνουμε ουσιαστικό έλεγχο και, τα, και είναι σύνηθες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος αυτό γιατί το ακούνε ακριβώς και από τους δικούς τους εθνικούς βουλευτές. Ας πούμε αυτό στην Γερμανία δεν ισχύει. Έχουν υπάρξει κάποιες προσπάθειες, έχει, έχουν, ε, έχει πάει υπόθεση και σε γερμανικό δικαστήριο και μάλιστα το, ε, ευρωπαϊκό, το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας το έχει απορρίψει το αίτημα. Γιατί αυτό είναι δουλειά άλλων και δεν χρειάζεται να ε, γίνεται ας πούμε έλεγχος ή να λαμβάνεται η οποιαδήποτε ανάληψη ευθύνης για τον γενικό προϋπολογισμό αλλά δεν γίνεται να δημιουργούνται και υποψίες ότι ένα κομμάτι της, ε, ε, του γενικού προπολογισμού χρησιμοποιείται για να αυξηθούν οι μισθοί. Αυτά δεν μπορούν έτσι να ύπτανται χωρί να υπάρχει καμία απάντηση. Και βεβαίως ε, και το ανώτερο δικαστήριο, το οικονομικό δικαστήριο στην Γερμανία είπε ότι οι Γερμανοί ευρωβουλευτέ δεν είναι υποχρεωμένοι να δίνουν λογαριασμό ουσιαστικά αλλά αυτό συμβαίνει μόνο στη Γερμανία. Σε άλλε χώρε είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η ε, λογοδοσία. Και θέλω να πω ότι στις χώρες όπου και βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με τις πολιτιστικές διαφορές στις χώρες λοιπόν όπου η απόλυτη διαφάνεια ε, για, τις, ε, για τα καταβολικοπή ποσά των προεδρίων κτλ. Είναι συνηθισμένο γεγονός. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις ακόμα και στους ε, βοηθούς των συγκεκριμένων ευρωβουλευτών. Αλλά τώρα, αν τα δούμε όλα αυτά μαζί, αν δούμε δηλαδή τι γίνεται και ποια είναι η κριτική που έρχεται από το κάθε κράτος μέλος μας, θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση που δυστυχώς θα μας δυσκολεύσει πάρα πολύ τη δουλειά. Στο παρελθόν υπήρξε και εσωτερικέ εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές που όταν είπαμε ότι όταν μιλούμε για εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υπερασπιστούμε αυτό που διαθέτουμε για τους ευρωβουλευτές μας Βεβαίω πάντα είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε επικοδομητικέ προτάσεις για την μείωση βεβαίως των δαπανών, αλλά δεν θα καταλύσουμε τα πάντα πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπιχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια του χρόνου πάλι θα έρθουμε μπροστά σε εκλογές. Και πρέπει να δούμε πώς παρουσιάζονται στην Ευρώπη οι ευρωβουλευτές. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήσαμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη οι ευρωβουλευτές να παρουσιάσουν αυτή τη δουλειά που κάνουν ε, για τους πολίτες της Ευρώπης. Να τους την παρουσιάσουν να φτάσει αυτή η δουλειά και το αποτέλεσμα της στους πολίτες. Γι' αυτό πραγματικά χαιρετίζω τις προσπάθειες που γίνονται εδώ στο Κοινοβούλιο, ε, είτε, το, είτε μέσω του Policy Department, είτε οποιασδήποτε άλλες προσπάθειες γίνονται, να συμμετέχουν οι πολίτες, να ενημερωθούν οι πολίτες της Ευρώπης για το τι γίνεται στην, στο Κοινοβούλιο. Ε, είτε μέσω του Facebook, είτε μέσω του Twitter. Πολλοί ευρωβουλευτές έχουν ε, λογαριασμού στα, ε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε το Voxbox. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι να χρησιμοποιήσει ο Ευρωπαίος πολίτης όλα αυτά τα μέσα για να ενημερωθεί. Έχουμε και την τηλεόραση του Κοινοβουλίου, το Europal TV. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν έτσι ώστε να διευκολύνουμε και την, ε, ε, και τον, και την παρουσίαση των, ε, της εργασίας μας και να ενημερωθεί ο κόσμος πολύ καλύτερα, να βελτιωθεί δηλαδή η εικόνα μας οι, ε, πραγματικά οι ε, υπάλληλοι του Κοινοβουλίου έχουν ε, λειτουργήσει πάρα πολύ καλά και για τη δουλειά που κάνουμε και για το πώς τελικά δρούν όλες αυτές οι επιτροπές που δεν είναι και λίγες και για το πώς μπορεί να παρουσιαστεί καλύτερα η δουλειά τους. Κυρίως και στους πολίτες που ενδιαφέρονται. Και γιατί πολλοί πολίτες μπορούν και να μας βλέπουν και να μας ακούνε στο ίντερνετ ακριβώς λόγω της δυνατότητας που έχουμε να μεταδίδονται οι συνεδριάσεις μας live στο ίντερνετ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει άλλος που να έχει ζητήσει το λόγο. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο πάλι στην εισηγήτρια, ως πρόεδρος της Επιτροπής, θα ήθελα να θέσω έτσι μια σκέψη εδώ σε εσά, την οποία θα συζητήσουμε αύριο με τον πρόεδρο Σούλτς, γιατί ήταν άρρωστος και ε, αναβάλαμε την συνεδρίασή μας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σκόπιμο εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού μαζί με τους, ε, και μαζί με τους υπολείπους συναδέλφους βεβαίω από τις υπόλοιπες ε, επιτροπές να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο, ένα κοινό τόπο για το πώς βλέπουμε τα καθήκοντα των επιτροπών μας, ποια είναι τα τεχνικά μέσα που χρειαζόμαστε ώστε να είναι αποτελεσματική η δουλειά μα και να επικεντρωθούμε σε κενά, σε ελλείψεις που τα έχουμε συζητήσει βέβαια πολλές φορές και ίσως να μην χρειάζεται να συμπεριλαμβάνονται κάθε φορά σε κάθε ψήφισμα για, τον, για, τον, την απαλλαγή. Ας πούμε στις ε, καταποκοπή αποζημιώσεις πάντα το, το θέμα αυτό πάντα το συζητούμε. Να σας θυμίσω ότι στον ιστορικό ε, στο δημοσιονομικό κανονισμό έχουμε δώσει στα κρατημέλη την ε, ε, δυνατότητα και μέσω του, το, το αλλά και μέσω του, του Ταμείου Συνοχής να χρησιμοποιήσουν δυνατότητες διευκόλυνσης και όταν μιλούμε για καταποκοπή αποζημιώσεις ε, πρέπει να γίνεται ο σωστό έλεγχος ε, για να γίνεται και ο διαχωρισμό ανάλογα με τις ε, αποζημιώσεις που δίνονται γενικώ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το θέμα είναι καυτό και το συζητούμε, το ξανασυζητούμε. Καλό θα ήταν λοιπόν κάποια στιγμή όλοι στο Κοινοβούλιο να καταλήξουμε σε, μια, σε ένα κοινό τόπο και να, επικοινωθούμε στα βασικά, στα ουσιώδη ζητήματα. Προφανώς θα πρέπει να το ξαναδούμε και στο μέλλον, για το πώ δηλαδή μπορεί το ένα κοινοβούλιο να έχει την ίδια, έτσι, να έχει μια ισότητα όπλων με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο μπορεί να στραφεί στα κράτη-μέλη. Ας πούμε, το προσωπικό του Κοινοβουλίου, είτε στη βιβλιοθήκη, είτε στις γραμματείες, σε σχέση με κάποια εθνικά κοινοβούλια ή σε σχέση με το Κογκρέσο στη ΣΥΠΑ είναι αρκετά έτσι, ταπεινό. Και όταν θέλουμε να έχουμε και καλή νομοθετική διαχείριση, καλή νομοθεσία, ε, πρέπει να έχουμε μια ισότητα όπλων με το Κοινοβούλιο, με τις ε, κυβερνήσεις ας πούμε, που έχουμε να ελέγξουμε ή όταν ε, νομοθετούμε, συνομοθετούμε με το Συμβούλιο. Αυτό ήθελα να σας το αναφέρω. Θα μας απασχολήσει λοιπόν και σε ό,τι αφορά τα away days, γιατί και εκεί μιλούμε για την, ε, για την ποιότητα εργασίας των επιτροπών. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρξουν ίσως κάποιες προτάσεις ως προς αυτό για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις ε, συνεδριάσεις μας. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο κατευθείαν στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους. Θα μπορέσουμε να εξετάσουμε λεπτομερώς τις διάφορες τροπολογίες που θα υποβληθούν. Διαπιστώνω ότι η Europal TV είναι ένα θέμα που συχνά αναφύεται. Υπάρχουν διάφορες τοποθετήσεις. Σε αυτή την έκθεση γίνεται λόγος για μια μελέτη κόστους απόδοσης, διότι εδώ πρόκειται περιφεάς ζώνης δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Διότι καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι είναι πολύ απόμακρη από τα κράτη-μέλη δουλειά που κάνουμε εδώ. Απ' την άλλη χρειάζεται και έλεγχος του, Euro, του κόστους του Europal TV και πρέπει να βρούμε τη μέση λύση. Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε μια συνένεση, να συμφωνήσουμε οι πολιτικές ομάδες, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε κάτι που θα είναι αποτελεσματικό. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο Γκαρίγα όσον αφορά το σημείο 55 που αφορά τα κτίρια και τα διά προβλήματα. Διότι δεν πρόκειται περί πολύ παλαιών κτίριων δεν δικαιολογούνται τέτοια προβλήματα. Το συζητήσαμε αυτό ήδη με τη Γενική Διεύθυνση την Αρμόδια και με το Γενικό Γραμματέα αυτό είναι, ξεπερνάει και τα διάφορα νομικά πλαίσια όσον αφορά τις διεκδικήσεις που μπορούμε να έχουμε, τις αξιώσεις που μπορούμε να έχουμε. Σας ευχαριστώ για την βοήθειά σας. Πρέπει πράγματι να τονίσουμε αυτό το ζήτημα ανεξάρτητα από το νομικό πλαίσιο όπως έλεγα, διότι θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιμείνουμε από αυτού. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη του προϋπολογισμού μας και πώς γίνεται η εξακρίβωση των δαπανών, ο έλεγχος των δαπανών. Τι γίνεται λοιπόν με τις δαπάνες. Αυτό είναι ένα ζήτημα σημαντικό. Ξέρουμε ποια είναι τα έσοδα, ποια είναι τα έξοδα, ξέρουμε ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα και από τούδο και στο εξή θα υποστηρίξουμε ό,τι χρειάζεται για να επικρατήσει διαφάνεια. Α μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι σε αυτά τα θέματα ιδιαίτερα σε αυτή την δύσκολη οικονομική ε, περίοδο μπορούμε να καταλήξουμε σε αρνητική κατάσταση, σε αρνητική θέση όσον αφορά τις δραστηριότητές μας. Ευχαριστώ Εύα. Προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 26 Φεβρουαρίου, Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση για το σημείο και περνάμε στο επόμενο σημείο. Σημείο 5. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και των φορολογικών παραδείσων. Ο Μπάρτστας είναι ο εισηγητής. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ήταν η καθήλια αρμόδια. Να δώσω λοιπόν κατευθείαν το λόγο στον εισηγητή. Μπαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γνωμοδότηση για την αρμόδια Επιτροπή. Όντως, εμείς προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που είχαν στη διάθεσή μας διότι η Επιτροπή Εκών του Κοινοβουλίου θα ψηφίζει ήδη το Μάρτιο, άρα πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Δίνω έμφαση σε κάποια σημεία, 12 είναι αυτά. Ε, φυσικά μιλώντας για την έκταση της φοροαπάτης, φοροδιαφυγής, αλλά και άλλα σημεία ε, σε σχέση με την απάτη που γίνεται με το ΦΠΑ. Καταρχήν, υπογραμμίζω την έκταση αυτού του προβλήματος και έχουν γίνει μελέτες για την φοροδιαφυγή και φοροαπαφυγή Ε, η οποία είναι απίθανη σε έκταση, ξεπερνάει δηλαδή πολλές φορές και τους προπολογισμού ε, χωρών μελών. Αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους, τα ελλείμματα ε, των χωρών, τα ελλείμματα χωρών που έχουν ε, αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαν να ρυθμιστούν για πολλά χρόνια στη συνέχεια. Υπάρχει φυσικά το θέμα της τεχνολογικής φύσεως έχουν βρεθεί. Έχουν βρεθεί νέοι τρόποι από τους ε, παράνομους να μπορέσουν να κάνουν ε, αυτές τις ε, απάτες μέσω φορολογικών παραδείσων. Έχω δει κάποιες μελέτες που έχουν γίνει στις κάτω χώρες όπου λέγεται ότι υπάρχουν πολλές εταιρείε επιχειρήσεις που υπάρχουν μόνο σαν γραμματοκιβώτια, μια εικονική θα λέγαμε ε, έδρα και αυτές διακινούν τουλάχιστον 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η έκταση αυτού του προβλήματος. Ένα τρίτο σημείο που αφορά την Επιτροπή μας είναι το εξής, ότι ο, ο, έλεγχος έχει μια αρνητική επίπτωση όσον αφορά τους επιχειρηματίες ε, για τους αρμόδιους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ένα μεγάλο, μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής ε, γίνεται από μεγάλες επιχειρήσεις και αυτό δίνει ε, αρνητικά σινιάλα θα λέγαμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να, δημιουργείται δηλαδή ένα ε, κακό παράδειγμα. Και ίσως να έχουν την εντύπωση ότι και αυτές μπορούν να ακολουθήσουν σε αυτό το μονοπάτι. Κάτι άλλο τώρα, τέταρτο. Είπαμε συχνά στην Επιτροπή μας ότι οι μεγάλοι γίγαντες της καπνοβιομηχανίας πληρώνουν σημαντικά ποσά σύμφωνα με συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί. Και με το πνεύμα αυτών των συμφωνιών αυτά τα ποσά θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουμε για τον αγώνα κατά του καπνίσματος. Αλλά μόνο 10% πηγαίνουν στην Κομισιόν και τα 90% πηγαίνουν στις χώρες μέλη, οι οποίες όμως δεν τα χρησιμοποιούν αυτά για τον αγώνα κατά του καπνίσματος. Τα βάζουν στον προπολογισμό τους. Πέμπτο στοιχείο. Ε, για το ΦΠΑ. Ε, μόνο γι' αυτό μιλάω σε αυτό το σημείο. Τα αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά στον προπολογισμό των χωρών μελών, διότι μειώνεται τα έσοδα για τους προπολογισμού, αλλά έχει επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Διότι ένα μέρος του ΦΠΑ καταλήγει στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτή η απάτη ε, έχει μεγάλες και ολέθριες επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά. Και δεν υπάρχει, θα λέγαμε, ε, ε, σωστός ανταγωνισμός. Τώρα, το ΦΠΑ είναι ένα σημαντικό μέρος ε, των δημοσίων εσόδων, περίπου 21% κατά μελέτες που έχουν γίνει. Αλλά αυτό το σύστημα οδηγεί και σε, κάποιες, σε κάποια κόστη. Τώρα, στο σημείο 7 αναφέρεται ότι όλα τα, τα συστήματα που έχουν να κάνουν με τη συλλογή του ΦΠΑ δεν έχουν αλλάξει από πολύ παλιά. Παρόλο, παρόλο που η οικονομία έχει αλλάξει. Άρα, τι γίνεται. Το, το μοντέλο συλλογής ΦΠΑ δεν ανταποκρίνεται στις δικές σημερινές δαπάνες. Όγδο στοιχείο. Το απευθύνομαι στο Συμβούλιο. Εδώ και χρόνια ε, έχουν ε, στο, στο τραπέζι τους ε, οδηγίες

Ίσως υπάρχει το θέμα μιας συνεργασίας ανάμεσα στα σύστηματα. Αλλά δεν μόνο αυτά, θα πρέπει να δούμε και τα θέματα των συνόρων, των τελωνίων. Δηλαδή χρειάζεται μια ανταλλαγή πληροφοριών. Διότι αν δεν γίνει, γίνεται κάτι τέτοιο, ε, διευκολύνεται η απάτη. Κάνω μια σαφή αναφορά σε αυτό και λυπάμαι που πολλές υπηρεσίες φορο... εφορίες στις χώρες μέλη δεν έχουν δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία, σε δεδομένα για να μπορέσουν να δουλέψουν. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μόνο ε, διαβρώνεται θα λέγαμε το σύστημα και αποδυναμώνεται. Επόμενο σημείο τώρα. Ο, ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοραπευγής πρέπει να γίνεται στα πλαίσια μιας ε, θα λέγαμε έκτασης τέτοια που να είναι αποτελεσματική. Οι έρευνες είναι δύσκολες, είναι χρονοβόρες και πολύ συχνά οι αρμόδιοι, οι υπάλληλοι που οι οποίοι έχουν δουλέψει πάνω σε αυτά τα θέματα κάνουν έναν αγώνα δεχομένως βρίσκονται κάποιοι υπεύθυνοι, αλλά οι ποινές είναι πολύ χαμηλές. Ε, και γίνονται και πολλές ατασαλίες. Άρα θα πρέπει να γίνει κατανοητό και αυτοί θα πρέπει να, πάρουν, ε, να αναλάβουν δηλαδή, τις ευθύνες τους και να είναι πιο σοβαροί με το έργο τους. Επίσης το θέμα της, ε, του ψηφιακού τρόπου δράσης ε, ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχουμε, πετύχουμε μια καλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα φορολογικά θέματα. Θα πρέπει να το ενισχύσουμε αυτό το θέμα. Αυτό το λέω στο 11, στο δυσμείο 11 και 12 το τέλος ε, είναι ένα σημείο το οποίο απευθύνεται στις χώρες μέλης και στην Επιτροπή ε, και έχει να κάνει ε, με τον ε, εξυγχρονισμό υπάρχει μια σειρά γνωμοδοτήσεων που απευθύνονται στην Επιτροπή Εκών του Κοινοβουλίου μας. Τα, τα πράγματα δεν γίνονται όπως έπρεπε. Λυπούμαστε γι' αυτό, το λέμε σαφέστατα στο τελευταίο σημείο, στη γνωμοδότησή μου. Ε, λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Ε, 26 Γενάρη είναι προθεσμία κατάσταση απολογιών. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε για να περάσουμε στην αρμόδια επιτροπή. Φυσικά τώρα είμαι στη διάθεσή σας για όποιες παρατηρήσεις έχετε να κάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να καλωσορίσω και τους εκπροσώπους της Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση Ταξούντο, ο κύριος Ραπώνη, και από τη Γενική Διεύθυνση Budget, ο κύριος Γκίλισε, από την Όλαφ, εδώ είναι ο κύριος ΜακΜάικλ. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Να δώσω τους λόγους, να, το λόγο τώρα στους συναδέλφους που έχουν ερωτήματα και για την Κομισιόν και για την Όλαφ, ε, πριν δώσω βεβαίω στους εκπροσώπους τη δυνατότητα να απαντήσουν. Ο κύριος Ρούμπιχ έχει πρώτο το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή γιατί πραγματικά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, πολύ ακριβή εργασία στην ε, Ευρώπη, τις, ευρωπα... επιχειρήσει, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, έχουμε επιβαρύνει πάρα πολύ. Και ουσιαστικά συμβάλλουν κατά 50% στο ΕΠ. Απασχολούν πάρα πολλού εργαζόμενου σε όλη την Ευρώπη και πληρώνουν και το 80% των φόρων. Επομένω κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι δίκαιο, ότι είναι σωστό οι μικρέ και οι ε, οικογενειακέ επιχειρήσει να επιβαρύνονται τόσο πολύ, τόσο δυσανάλογα. Για τις μεγάλες, τις διεθνείς επιχειρήσεις, ε, ε, είμαστε πιο ε, έτσι, ε, δεν είμαστε τόσο αυστηροί και αυτό δεν είναι σωστό. Το ερώτημα μου είναι, έχει γίνει κάποια σκέψη για τον φορό συναλλαγών, για τις διασυνοριακές δραστηριότητε, ίσως να ληφθούν υπόψη, θα μπορούσε ίσως αυτό να αποτελέσει ένα, έτσι, μια εργασία σημαντική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει σκεφτεί κάποιος κάτι επ' αυτού. Και επίσης, αυτός ο φόρος συναλλαγών, κυρίως για, τα, για τις μικροπιστώσεις θα μπορούσε να εφαρμοστεί, για να δοθεί δηλαδή ένα κίνητρο για α, φοροελάφρυνση. Να υπάρξει δηλαδή μια ισορροπία στο σύστημα. Νομίζω ότι η Σλοβακία μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα υποδειγματικό μοντέλο ως προς αυτό για την ε, ανάπτυξη, για, νέες, ε, για την ε, απασχόληση και για θέσεις εργασίας. Και πάντα ήταν πολύ αυστηρή απέναντι στους φορολογικού παραδείσους και νομίζω ότι έχει λειτουργήσει πολύ καλά το πρόγραμμά τη. Ευχαριστώ βεβαίω και την Κομισιόν που μελετά το θέμα για τον τομέα αυτό και για το πώ δηλαδή στο μέλλον θα μπορέσουμε να έχουμε μια αλφα ισορροπία στο σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπιχ. Ο κύριο Ντεγιόγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Στάς, τον εισηγητή. Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο σε μια γνωμοδότηση να, όταν έχουμε την έκταση ενός τέτοιου θέματος ε, και περίπλοκο μάλιστα. Πώς μπορεί κανείς να κάνει το καλύτερο τώρα. Όπως και να έχει το θέμα, θα προσπαθήσω να καταθέσω μια σειρά ε, τροπολογιών στο πνεύμα του εισηγητή. Καταρχήν, μία παρατήρηση. Στην αγγλική εκδοχή που έχω στα χέρια μου, που, η μόνη που βρήκα, μιλάει, μιλάνε, αναφέρεται tax evasion. Ε, υπάρχει το θέμα μεταξύ tax evasion tax avoidance. Είναι διαφορετική όρη. και ότι θα χρειάζονται 8 ε, χρόνια για να μπορέσει κανείς, ε, για 8 χρόνια θα μπορέσει κανείς να καλύψει τις δαπάνες με τα χρήματα της, ε, της φοροαπάτης. Τώρα, κάτι άλλο. Σίγουρα. Είναι λογικό να πληρώνει κανείς τους φόρους του εκεί που γίνει, έχει τη δραστηριότητά του. Αλλά αυτό στην πράξη δεν ισχύει. Δεν εφαρμόζεται. Η αρχή δεν ισχύει παντού και πολλές φορές γίνονται διάφορα προβλήματα. Ε, πληρώνει κανείς φόρο σύμφωνα με κάποιες συνθήκες που ισχύουν. Πολλές φορές δεν πληρώνεται κανένας φόρος. για μένα οι, ε, οι συνθήκες που ισχύουν για, για τους φόρους είναι πολύ σημαντικές και αναφέρονται και κάτω χώρες. Και αυτό ισχύει διότι οι κάτω χώρες έχουν πολλές ε, συμβάσεις με διάφορες χώρες. Ορισμένες από αυτές τις χώρες έτσι αμφίβολες θα λέγαμε ε, καταστάσεως. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε προσοχή πάνω σε αυτό το θέμα. Στη συνέχεια υπάρχει η έκθεση του ΟΣΑ που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, αναφερθήκαν σε αυτό το θέμα υπάρχει μια, ένας κατάλογος που παρουσιάζεται με πολύ καλές ιδέες θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά σε αυτήν τον κατάλογο δράσεως που μας προτείνει ο ΣΑ επίσης για τις κυρώσεις επιχειρήσεις που έχουν κάνει κάτι τέτοιο με φοροαποφυγή θα πρέπει να έχουν κάποιες χειρώσεις. Θα πρέπει να ισχύσουν τα όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά, τη στιγμή που έχουμε 28 διαφορετικά μοντέλα όσον αφορά τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, καταλαβαίνετε αν μπορούσε να υπάρχει μια συγκρισιμότητα θα, υπήρχε και θα είχε μειωθεί και αυτή η φοροαπάτη. Για μένα είναι μια καλή γνωμοδότηση, η στόχη είναι σαφέστατη και θα πρέπει να δώσουμε φόρμα σε αυτούς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάννη έχει το λόγο. Γιάννη eh, Κοιτάξτε, φαίνεται ότι τα Ολλανδικά είναι η lingua franca. Θα μιλήσω λοιπόν τη μητρική μου γλώσσα. Όσον αφορά τα συμπέρασματα του κειμένου είναι πολύ καλά, αλλά θα να αναφερθώ στο, στο φορολογικό παράδοσο Ολλανδία. Ο τίτλος του, της εκθέσεως είναι «Καταπολέμηση της απάτης, της φοροδιαφυγής και, και καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων». Δεν νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί η Ολλανδία δεν έχει εγκληματική συμπεριφορά ή όχι. Ε, αν είναι ικανοποιητική κατάσταση ή δεν είναι, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ε, θα πρέπει να έχουμε ειδική επιτροπή ερευνητική που θα έπρεπε να το εξετάσει από την κάτω βουλή. Αλλά δεν νομίζω ότι παραβιάζονται οι νόμοι στην Ολλανδία. Βέβαια ζούμε σε δημοκρατίες, ε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε τις φοροαπάτες σε τέτοια κλίμακα. Και δεν μπορώ να φανταστώ τι συμβαίνει πραγματικά αυτό. Στο 90%, το 90% των χρημάτων των καπνοβιομηχανιών που εικάζεται ότι πηγαίνουν στα κράτη-μέλη δεν είμαι σίγουρος αν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να θεωρήσουμε τις συμφωνίες που υπάρχουν. Στα πλαίσια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου όλοι μιλάνε για οικονομίες. Αυτή είναι μια μορφή ε, φόρου ε, που ε, και οι πόροι πηγαίνουν στα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω πόσο παλιά είναι η συμφωνία αυτή που υπάρχει. Θα πρέπει ίσως να εξεταστούν οι λεπτομέρειες και να δούμε μήπως στην Ευρώπη μπορούμε να πάρουμε περισσότερα από τα 10% που αναφέρονται και μήπως μπορούμε να πάρουμε κάτι παραπάνω από κενές υποσχέσεις για να χρησιμοποιηθούν και τα χρήματα τα υπόλοιπα των 90% στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ Γιάννη. Ο κύριος Ροντή έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας. Είναι ένα θέμα το οποίο επεξεργάζεται τακτικά. Ευχαριστώ για αυτή την έκθεση. Έχω τρεις σκέψεις να εκφράσω. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τη διεθνή απάτη, μετά από διάφορε ενδιάσει του G20, όσο πιο ανοιγόμαστε προ την παγκοσμιοποίηση, τόσο αυξάνεται η μεγάλη διεθνή απάτη. Και διαρωτώ με ποια θα μπορούσε να είναι η συνεισφορά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω με του υπαλλήλου μα, με τα συστήματα που έχουμε πληροφορική και ενημέρωση, πώ μπορούμε εμεί να συμβάλλουμε, να βάλουμε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια που γίνεται για την καταπολέμηση της διεθνούς απάτης, που γίνεται πραγματικά προβληματική. Υπάρχει σόρευση σημαντική κεφαλαίων σε κάποιους τόπους στον πλανήτη και μετά να κυκλώνονται οι πόροι σε παράνομες δραστηριότητε. Θα πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί. Διερωτώ με, μήπως πρέπει να κάνουμε κάποια παράγραφο, κάποια ε, τροπολογία. Στη συνθήκη την εμπορική που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις διμερείς συμφωνίες να μπορούμε να, έσουμε, να έχουμε κεφάλαια που αφορούν τη συνεργασία στο θέμα της ε, απάτης κάθε φύσης, κάθε είδους κυρίως ε, σε θέματα φορολογικά. Αυτό αφορά τους φορολογικούς παραδείσους, ε, αφορά όλα όσα άπτονται της διεθνούς φορολογικής απάτης. Δεύτερον, στην έκθεση, Μπάρτ, δεν αναφέρεται κάτι, είχα διαβάσει τον τύπο ότι είχα διαπιστωθεί απάτες όσον αφορά το σύστημα ανταλλαγής ποσοστώσεων διοξιδίου του άνθρακος. Είναι πάντα επίκαιρο αυτό. Μήπω πρέπει να γράψουμε μία παράγραφο όσον αφορά αυτού του είδου ε, την απάτη, αν υφίσταται και ποια είναι τα αποτελέσματα τη προσπάθειας καταπολέμησης αυτού του είδου τη απάτες. Μετά στην παράγραφο 9 και στην παράγραφο 12 γίνεται αναφορά στα τελωνία. Γίνονται εκθέσει, γίνονται επισκέψει, το ελεκτικό συνέθριο μα υποβάλλει εκθέσεις και βλέπουμε ότι έχουμε τελωνιακό σύστημα που είναι πολύ ατέλες. Υπενθυμίζω όμω ότι τα τελωνία είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε, δεν έχουμε και πολλέ αρμοδιότητε. Έχουμε τη Γεωργία, έχουμε τα Τελωνία. Ήμουν εισηγητή εδώ και πολλά χρόνια για μια έκθεση για τη σχέση τη ποιότητα του τελωνιακού συστήματο με το διεθνέ εμπόριο. Και είχαμε εντοπίσει και είχαμε διαπιστώσει ότι επρόκειτο περί προβλήματο. Είχα προτείνει τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα οι ε, ε, τελωνιακοί δημόσιοι υπάλληλοι να είναι υπό την εξουσία τελωνιακή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε μου είπαν όχι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε κλπ. και Μα τι λέτε, οι υπουργοί είπαν ότι δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε για κάτι τέτοιο. Δεν θα κόστιζε περισσότερα χρήματα, αλλά έτσι θα είχαμε μία αρχή που θα ήταν ευρωπαϊκή αρχή, ευρωπαϊκή υπηρεσία. Και είχα προτείνει να διεξαχθεί τουλάχιστον μία μελέτη. Μήπω μπορούμε να επαναπροβάλλουμε αυτή την ε, ιδέα να γίνει με μελέτη στον μεσοπρόθεσμα, να δούμε να, είναι, ε, να ενταχθούν στο δημόσιο τομέα τελωνιακή, να δημιουργήσουμε Ευρωπαϊκή Αρχή Τελωνίων. Έτσι να αποφύγουμε το παρόν σύστημα, όπου είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα μεν, αλλά ανατίθεται στα κράτη-μέλη η αρμοδιότητα. Και διαφέρουν οι ιδιότητες των τελωνίων στα σύνορα, κυρίως στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα με απάτες, προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, προβλήματα όσον αφορά τον, ε, το σεβασμό των διαφόρων εμπορικών συνθήκων κλπ. Ξαναθέτω αυτή την ιδέα, την ξαναρίχνω. Δεν ξέρω μήπως θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε μια έκθεση αυτού του είδους. Ευχαριστώ. Επόμενη η κυρία Μακόβα. Ευχαριστώ. Το 2011 η γκρίζα οικονομία ήταν 90% του ΑΕΠ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 2,4 ε, δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Δεκάδες δισεκατομμύρια μένουν σε υπεράκτιους τόπους και δεν φορολογούνται. Η απάτη του ΦΠΑ μειώνει τα έσοδα των κρατών μελών και επηρεάζει και τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή διότι είναι ουσιαστική πηγή εσόδων των ίδιων πόρων ο ΦΠΑ. Και η φοραπάτη υπονομεύει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και εμποδίζει και τον θεμητό ανταγωνισμό. Η καταπολέμηση της φοραπάτης και φοροδιαφυγής θα πρέπει να εστιάζεται επί πέντε κατευθύνσεων, αξώνων. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βελτιώσουμε την τρόπο συλλογής των ίσπραξης των φορών, δεν θα επισέλθω στις λεπτομέρειες αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιωθεί ή να αλλάξει ριζικά σε κάποια κράτη-μέλη. Υπάρχουν κράτη-μέλη στα οποία η ίσπραξη των φόρων είναι αποδίδει κάτω από 10%. Μετά, χρειάζεται διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, των φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Είναι κάτι που πρέπει να ενισχυθεί και να βελτιωθεί. Και διασυνοριακή συνεργασία με τις χώρες εταίρους χρειάζεται, χώρες που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εδώ πρόκειται περί χρημάτων που περνάνε τα σύνορα σε δευτερόλεπτα και θα πρέπει να συνεργαστούμε. Επί της αρχής ακολουθήστε τα χρήματα και πέρα από τα σύνορα. Όποια και να τα σύνορα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όσον αφορά λοιπόν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έχω ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δρομολογήσει εξολόγηση αντιχτύπου όσον αφορά ε, συριακό αριθμό εντοπισμού φορολογικού και αν ναι, ε, ποια είναι τα αποτελέσματα προς το Συμβούλιο. Το Ελεκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότειναν ε, να διενεργηθεί έρευνα όσον αφορά την καταβολή του ΦΠΑ στις χώρες προορισμού να ελέγχετε τι γίνεται με την καταβολή του ΦΠΑ στα και κάτι μέλη. Πότε θα συνεχιστούν οι συζητήσει στο Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Άλλο. Χρειαζόμαστε εργαλεία. Εργαλεία για να αντιμετωπιστούν όλες οι μέθοδοι φόρο διαφυγής και απάτης. Παράδειγμα. Ιούνιος 2008. Με Δεκέμβριο 2009 5 δις ευρώ χάθηκαν λόγω απάτης ΦΠΑ όσον αφορά τις, ε, τα ποσοστά εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος. Στην προηγούμενη Ολομέλεια, μετά τη ψηφοφορία για την έκθεση Κάσα, καλωσόρισα την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργηθεί μηχανισμό ταχεία αντίδραση. Λυπούμε ότι η οδηγία έχει μπλοκάριστεί ακόμα στο Συμβούλιο. Άλλα ερώτηση απευθύνω στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο πότε προτίθεται να προχωρήσει για το μηχανισμό γρήγορης αντίδρασης και τη σχετική οδηγία. Τέλος, ο περίπλοκος χαρακτήρας νομοθεσίας για το ΦΠΑ, όπως και στις δημόσιες προμήθειες. Πρέπει να πω ότι η νομοθεσία είναι περίπλοκη και επαχθής είναι πανεύκολο να βρει κανείς παραθυράκια για να ξεφύγει και να διαπράξει απάτη και να φοροδιαφύγει. Σαφής, απλή, διαφανής νομοθεσία είναι η εγγύηση ότι θα εφαρμόζεται ο νόμος και θα μειωθούν οι δυνατότητες απάτης. Αυτά. Εκτιμώ την έκθεση του εισηγητού και όπως οι προλαλήσατε συνάδελφοι και εγώ πιστεύω ότι παρόμοια είναι η προσέγγισή μας και ελπίζω στο τέλος να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ο επόμενος. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή. Έξοχη έκθεση του. Είμαι ο εισηγητής για την έκθεση ΠΙΦ φέτος. Υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ αυτής εκθέσεως και του δικού μου θέματος. Κυρίως το θέμα της απάτης ΦΠΑ. Και κυρίως όσον αφορά το καπνό, τα προϊόντα καπνού και τα σιγαρέτα. Η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού θα πάει στο Καλίνιγκρα σε μερικούς μήνες για να εξετάσει την κατάσταση. Έγινε ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή αυτή. Συζητήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ινόλαφ για το σοβαρό αυτό θέμα. Κάτι με εξέπληξε από την ανταλλαγή απόψεων. Δηλαδή κάθε κράτος μέλο χρησιμοποιεί διαφορετικά συστήματα και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Τα κράτη-μέλη τώρα πλέον γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτά. Αλλά υπάρχουν διαφορέ με τον τρόπο χρήση των συστημάτων ελέγχου, με τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλουν τα μέτρα κατά πολέμηση απάτη και με τον τρόπο που επιβάλλουν τι κυρώσει. Το είπατε κι εσεί, νομίζω, όταν μιλήσατε. Ένα ερώτημα περισσότερο προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι γίνεται ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν ομοιόμορφη προσέγγιση όσον αφορά τους ελέγχους, επιβολή των νόμων και την επιβολή κυρώσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κυλακάκης έχει το λόγο. Ε, thank you. Ε, I would like to... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω αναφερόμενος Ε, sorry. Ε, ο Mr. Για την πρόταση του κυρίου Οντί, ε, για το θέμα των τελωνίων. Στο θέμα των τελωνίων προκύπτει με μεγάλη σαφήνεια από έρευνες που έχει κάνει η Διεθνής Διαφάνεια ότι υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά στις τελωνιακές αρχές. Η διαφθορά αυτή είναι πανευρωπαϊκή, ε, ιδίω αν υπολογίσουμε ότι πολλά από τα σύνορα της Ευρώπης όπου υπάρχουν τελωνία είναι χώρες που έχουν κακή βαθμολόγηση σε ό,τι αφορά τους δείκτες της διεθνούς διαφάνειας. Οπότε η σκέψη του κυρίου Οντί, του συναδέλφου, ότι θα μπορούσαμε να οθήσουμε σε μια πολύ πιο ευρωπαϊκή ε, πολιτική, έναν έλεγχο ευρωπαϊκό των τελωνιακών αρχών, ε, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και θα μπορούσαμε να πάμε και σε μια ενδιάμεση πρόταση κατά την οποία η, αν μη τι άλλο ε, να υπάρχει τουλάχιστον μια ισχυρή ευρωπαϊκή αρχή ελέγχου αυτών των υποθέσεων. Διότι στην πραγματικότητα, αν δείτε, ο Όλαφ συνολικά έχει κάνει τα τελευταία ε, πέντε χρόνια ε, κάπου, αν θυμάμαι καλά, 600 ε, συνολικά, 600-700 έρευνες, investigations και από αυτές μόλις οι 300 είχαν κάποια συνέχεια. Και αυτό αφορά το σύνολο των ε, ευρωπαϊκών υποθέσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι χρειαζόμαστε πολύ ισχυρότερη παρέμβαση σε αυτόν τον τομέα. Και θα τελειώσω δίνοντας έναν αριθμό μόνο. Με βάση τα στοιχεία που ε, παρουσίασα στην έκθεση την ειδική που έκανα για την διαφθορά στη, δημόσια διοίκηση των κρατών μελών, κάθε χρόνο γίνονται μικροδωροδοκίες ε, στα τελωνία της Ευρώπης ε, περίπου 600.000. 600.000 μικροδωροδοκίες. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ, συνάδελφε Σκυλακάκη. Να δώσουμε κατευθείαν το λόγο στην Κομισιόν. Έχουν τεθεί κάποια ερωτήματα ποιον, ε, σε ποιον να δώσω το λόγο, ποιος θα απαντήσει. Κάποιος από την Κομισιόν, ο κύριος Ραπώνη, ο κύριος Κίλησε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω όσον αφορά τα θέματα φορολογικά. Θα πρέπει να γίνει μια διάκριση Μέσα στην φόρα και ε, με την άλλη απάτη, διότι χρησιμοποιεί κανείς νόμιμα μέσα για να μειώσει το φόρο. Ενώ είναι άλλη μορφή απάτη φοροδιαφυγή. Παρόλο που ηθικά η φόρα απαφυγή είναι καταδικαστέα, όπω ε, όπως γνωστόν, ε, γνωστό μιλάμε για tax planning. Εδώ ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα όσον αφορά αυτή τη δραστηριότητα. Έχουμε το εθνικό επίπεδο, όπου εδώ οι αρμοδιότητε είναι των εθνικών αρχών για να κάνουν τον αγώνα κατά τη Έχουμε το ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ, εδώ έχουμε να κάνουμε τη συνεργασία ανάμεσα σε χώρες μέλη. Αυτή η συνεργασία θεωρούμε στην Επιτροπή ε, ότι υπάρχουν τα νομικά μέσα, αλλά είναι χώρες μέλη που δεν χρησιμοποιούν αρκετά αυτά τα μέσα που υπάρχουν ε, τα νομικά και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ε, θα πρέπει κανείς να απευθυνθεί περισσότερο στις χώρες μέλη. Μετά έχουμε τη διεθνή διάσταση, δηλαδή πέρα από τα όρια της ευρωπαϊκής επικράτειας. Και εδώ έχουμε να κάνουμε τη συνεργασία τη διεθνή, που είναι σημαντική. Έχουν αναφερθεί παραδείγματα, Φερρυπίν, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει διαπραγματεύσεις εμπορικής φύσεως, εμείς πάντοτε ζητάμε να υπάρξει ένα κεφάλαιο που έχει να κάνει με την φορολογική διαφάνεια. Αυτό λειτουργεί με κάποιες χώρες, όχι με κάποιες άλλες, οι οποίες αρνούνται να εντάξουν ένα τέτοιο κεφάλαιο σε, σε μια συνθήκη εμπορική, σύμβαση εμπορική. Σε διεθνές επίπεδο ε, έχουμε κυρίως διμερεί συνεργασίες, συμβάσεις ανάμεσα σε χώρες, μια τρίτη χώρα με μια ευρωπαϊκή φερρυπίνη. Μήπως τώρα εδώ κανείς αναρωτιέται ότι θα ήταν καλύτερα να έχουμε σε διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια τρίτη χώρα. Αυτό προσπαθούμε να ζητήσουμε εδώ και χρόνια το ζητούμε από τι χώρε μέλη. Όσον αφορά το ΦΠΑ, εμείς προβληματιζόμαστε εδώ και καιρό να ζητήσουμε εντολή από το Συμβούλιο του ώστε η Επιτροπή να κάνει διαπραγματεύσει για μια ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά το ΦΠΑ. Ξέρετε, ε, κυρίως αυτό αφορούσε ε, προϊόντα εμπορικά ε, προϊόντα. Τώρα όμως έχουμε υπηρεσίε. και είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να ελέγξει τη, ε, δραστηριότητα αυτή. Έχουμε τις επικοινωνίε. Φέλπιν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια διεθνή ενισχυμένη συνεργασία και θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι, τους διεθνείς εταίρους της. Ε, τα την ομάδα των 20 που είχαμε συζητήσει. Εδώ αναφερθήκαμε στο tax planning. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ε, υπάρχουν συμβάσεις δι, διμερείς. Όταν είπαμε για την αφο, απάτη στο ΦΠΑ και για την, το διοξίδιο του άνθρακος, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μια μείωση αυτής της απάτης, αλλά έχουν περάσει άλλα προϊόντα. Το φυσικό αέριο πίνο Και στην ηλεκτρική ενέργεια. Γι' αυτό η Επιτροπή έχει καταθέσει μια πρόταση για μηχανισμούς γρήγορης δράσης, ούτως ώστε να υπάρξει μια νομική βάση η οποία θα επιτρέψει στις χώρες μέλη να μπορέσουν καλύτερα ε, να δράσουν ξαφνικά αν αυτό χρειαστεί. Για το διεξίδιο του άνθρακός έχει πληρώσει μια χώρα 3 δισεκατομμύρια σε δύο μήνες ε, θα πρέπει να είναι κανείς γρήγορος στον αγώνα κατά της απάτης. Τώρα, για τις κυρώσεις, ακόμα και φορολογικές, η Επιτροπή ζήτησε από τις χώρες μέλη να δουλέψουν πάνω σε αυτό, αλλά οι χώρες εν γέννη αρνηθήκανε. Λέγοντας ότι οι ποινικέ και άλλες ε, κυρώσεις έχουν να κάνουν με ε, το νομικό δίκαιο και δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο αυτό το θέμα. Όσο για την φορολογία των της μεταφοράς κεφαλαίων. Ξέρουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε και ένα θέμα αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εφαρμογή αυτού του φόρου δεν θα πρέπει να, τις, να ισχύει για αυτές. Επίσης, για ένα άλλο θέμα στο οποίο δεν έχουμε κάνει ε, μελέτη για μια δράση και θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω συζητήσει με τι χώρες μέλη πριν να προχωρήσουμε σε μια αξιολόγηση ε, και για το θέμα που έχει να κάνει με αυτό το νούμερο ε, θα λέγαμε ταυτοποίηση όσον αφορά το ΦΠΑ. Να πω τώρα προς ενημέρωση ότι το River Chart, το και θέμα αυτό που έχει να συζητηθεί με το ΕΚΟΦΗΝ στην επόμενη φορά, τέλη Μαρτίου, και το Συμβούλιο έχει μεγάλη πλειοψηφία ε, που δείχνει ότι οι περισσότερε χώρες είναι υπέρ, τρει-τέσσερι είναι κατά για άλλου λόγου και είναι ένα θέμα το οποίο όμω έχει να κάνει με την ομοφωνία. Mm. Ωραία. Να δώσω το λόγο και στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού για τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Παρακαλώ αν θέλετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση ήταν αρκετά πλήρης. Εγώ δεν έχω πολλά να προσθέσω σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες. Μιλούμε για το ΦΠΑ που είναι η βάση για τα έσοδα. Αν δούμε το σημείο 5, βλέπω ότι είναι πολύ το σωστό αυτό που περιλαμβάνει. Ε, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που γράφει εκεί. Και πρέπει να πω ότι η απάτη με το ΦΠΑ ε, έχει πραγματικά σημαντικές ε, συνέπειες στα έσοδα που προκύπτουν από τον ΦΠΑ. Και βεβαίω έχει και συνέπειε και στα κράτη-μέλη. Αν δούμε τι ε, συνέπειε που έχει στα κράτη-μέλη, είναι τελείω διαφορετική η κλίμακα. Α πούμε, όταν η απάτη περιλαμβάνει 100 ευρώ και ας πούμε δύο κράτη-μέλη, οι συνέπειες που θα έχει ε, έχουν να κάνουν με το ποιο είναι το κράτος στο οποίο έγινε η απάτη. Δηλαδή, εγώ ζω εδώ, α πούμε στην Ολλανδία. Α πάρουμε το Βέλγιο και την Ολλανδία. Αν μιλούμε για μια απάτη 100 ευρώ, τότε οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκό, στον ευρωπαϊκό ε, προϋπολογισμό, αν η, αν απάτη γίνει στο Βέλγιο, τότε 98-50 είναι οι επιπτώσεις στο Βέλγιο και για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι το 1,5 ευρώ που απομένει. Αν η απάτη γίνει στις κατοχώρες, τότε οι επιπτώσεις είναι 75 λεπτά για τον, ε, ε, για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και αυτό που λέει ο κύριος Στάς στο σημείο 5 είναι απολύτως σωστό, μόνο αυτό που λέει είναι σαν να υπονοεί ότι είναι παρόμοιες σε συνέπειες. Και εκεί, αν μπορούσα να κάνω μια πρόταση, θα ήθελα να υπάρξει μια αλφα απόχρωση, γιατί ο, ο, ο φορολογούμενος που θα το διαβάσει θα θεωρήσει ότι, μάλλον θα έχει μια τελείως διαφορετική εντύπωση από αυτή που όντως ισχύει με βάση τούτη την παράγραφο. Α, κατά τα λοιπά δεν έχω άλλες παρατηρήσεις να κάνω. Ωραία. Περνάει και η ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ σύντομε παρατηρήσεις σας. υπήρξε ένα ερώτημα για την Όλαφ. Παρακαλώ να δώσουμε το λόγο στην Όλαφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, από τη Γενική Διεύθυνση Budget είμαι για, τις, ε, για τους ίδιους πόρους. Να... Ένα σημείο μόνο θέλω να θίξω. Σε σχέση με το σημείο 7 που λέει ότι, ότι το μοντέλο συλλογής ε, ΦΠΑ δεν έχει αλλάξει και επομένως οδηγεί σε σημαντικά σε σημαντικές απώλειες για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ο ΦΠΑ ε, ε, ε, ε, ουσιαστικά περιλαμβάνεται και στην τιμή που έχει το κάθε προϊόν. Και επίσης να πω ότι η Γενική Διεύθυνση Budget κάνει τακτικούς ελέγχους των, ε, των ε, πόρων και δίνει ιδιαίτερη σημασία στους τελωνιακούς ελέγχους που κάνουν τα κράτη-μέλη. Ελέγχει τι δράσεις που αναλαμβάνουν σε ό,τι αφορά την ε, διεξαγωγή των ε, ε, ελέγχων και αξιολογεί βεβαίω και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων. Επιπλέον, πέραν των ελέγχων που κάνει, παρουσιάζει κάποιε θεματικέ εκθέσει για, διάφορα, για διάφορα θέματα για του τελωνικού ελέγχου στα κράτη-μέλη στη Συμβουλευτική Επιτροπή για τους ίδιους πόρους και στην ομάδα για την Αταλονική Πολιτική. Ας πούμε, το 2011 παρουσίασε μια θεματική έκθεση για τη στρατηγική για τους τελωνικούς ελέγχους, το 2012 θεματική έκθεση για, τις, ε, ε, για τους εκτελονισμούς και όλα αυτά γίνονται για να τονιστούν τομεί όπου θα μπορούσαν όντω να ε, ενισχυθούν οι τελωνιακοί έλεγχοι που κάνουν τα κράτη-μέλη ω προ αυτού του τομεί. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να δώσουμε τον λόγο στον Κέβιν Μακμάικολ από την Όλαφ. Υπήρξαν δύο ερωτήματα προς την Όλαφ. Παρακαλώ, αν θέλετε να μας απαντήσετε για τον ρόλο της Όλαφ σε σχέση με τα ερωτήματα που σας έθεσαν ή θα μπορούσατε και γραπτός να μας υποστείλετε την, την απάντησή σας, όπως θέλετε. Μπορώ να απαντήσω στο εξή. Όταν λήξει η πρώτη συμφωνία για τα πρώτα καπνού, Philip Morris International το 2016. Οι άλλε λήγουν 20-22 και πιο πέρα. Η πρώτη δυνατότητα για να κάνουμε κάτι διαφορετικό θα είναι το τέλος του 2016. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε και πάλι το λόγο τώρα στον εισηγητή. Ε, να σας πω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών δεν είναι 26 Φεβρουαρίου, είναι η Δευτέρα, Τετάρτη η Δευτέρα 4 Μαρτίου. Συγγνώμη. Παρακαλώ, εισηγητή. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που παρατάθηκε η προθεσμία και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε χρόνο να ανισχύσουμε τη θέση μας. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Ε, ευχαριστώ τον κύριο Ρούμπιχ. Το κείμενο ε, που έχετε εκεί είναι ένα κείμενο για το οποίο δεν είχα γνώση. Καλή θα είναι να ξανασυναντηθούμε, να δούμε να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό. Οι παρατηρήσεις του κ. Ντεγιόγκ ήταν κατάλληλες, σωστές. Όπως έλεγα, ε, είναι μια σειρά περιορισμένων μέσων. Ίσως θα πρέπει να ξαναδώ το θέμα των τροπολογιών. Προστείνεται μια σειρά σημαντικών θεμάτων. Τώρα το evasion και avoidance, αυτοί οι δύο όροι, είναι στα αγγλικά. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε σωστά τα πράγματα. Αλλά ε, είχαμε δεχτεί κάποια πίεση. Για να δούμε πώς ακριβώς έχουν τώρα τα πράγματα. Η έκθεσή μου συνετάχθη πριν από τη δημοσίευση αυτή της έκθεσης. Θα ξαναδούμε λοιπόν αυτό το θέμα, θα το κοιτάξουμε μια τροπολογία. Σας το εγγυώμαι. Τα θέματα που σφίξατε είναι αποδεκτά. Τώρα για τις κάτω χώρες δεν ήθελα να πάρω ξανά το παράδειγμα των κάτω χωρών. Σίγουρα θα μπορέσουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το θέμα για το ε, του καπνού και είναι σωστέ και παρατηρήσεις όσον αφορά για το σύστημα το τελωνιακό. Ίσως να, να δούμε μεταξύ, με τους συντονιστές τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό το θέμα με την, τα τελωνία. Μήπως μια έκθεση πρωτοβουλίας. Αναφέρει και το θέμα του διοξίδιου τα ανθράκα. Απάντησε πάνω σε αυτό η Επιτροπή, η κυρία Μακοβέη, πρότεινε ένα πρόγραμμα ουσιαστικά δράσης για τη βελτίωση του συλλογής ε, ε, φόρων, τη συνεργασία, τη διασυνοριακή, ε, μια αξιολόγηση των επιπτώσεων. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούμε να το εντάξουμε αυτό το θέμα και επίσης να απευθύνουμε μια σειρά ερωτήσεων στο Συμβούλιο ο, για τον Σιώδη Συντηγητή συμφωνώ με αυτά που είπε. Υπάρχει εδώ πέρα μια σειρά θεμάτων που μας προβληματίζουν και σίγουρα θα συζητήσω μαζί σας πάνω, ε, πάνω σε αυτό και τον κύριο Σκυλακάκη ε, έχω λάβει υπόψη της παρατηρησού. Είμαι λοιπόν διαθέσιμος να συνεργαστώ με όλους. Μέχρι 4 Μαρτίου λοιπόν έχουμε περιθώρια και, και συνεχίζουμε στο δεύτερο ήμιση του Μαρτίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την γνωμοδότηση. Κλείνουμε το σημείο αυτό. Νομίζω ότι ο κύριο Στάσπρη πρέπει να πάει και σε άλλη συνεδρίαση, σε άλλη επιτροπή. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Ε, ακούσαμε κάποια εισαγωγικά σχόλια. Η υποβολή τροπολογιών για, αυτά, για αυτές τις υπηρεσίες είναι η 26 Φεβρουαρίου. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Ανδρέα Τσέσκοβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Φέτος, λοιπόν, μαζί με τον συνάδελφο Τσαρνιέσκι από την ομάδα μας μοιράσαμε τα καθήκοντά μας. Τα καθήκοντα που αφορούσαν την απαλλαγή για τους άλλους οργανισμούς, για τα άλλα θεσμικά όργανα. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του που απουσιάζει. Ε, ο συνάδελφος μου ζήτησε να διαβάσω τι έχει να πει ε, εκείνος, να μιλήσω εκ μέρους του. Ταυτόχρονα θα ήθελα να σας παρακαλέσω αν θα μπορούσα να αλλάξω την, ε, σειρά των διαφορετικών οργάνων, ούτως να μπορέσω να σχετίσω πρώτα απ' όλα τα δικά μου σχόλια, να τα παρουσιάσω και μετά να διαβάσω και τα σχόλια του συναδέλφου. Συμφωνείτε λοιπόν να αλλάξω τη σειρά. Αν συμφωνείτε μπορώ να συνεχίσω. Καλώς. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, στην προηγούμενη συνεδρίαση παρουσία εκπροσώπων άλλων θεσμικών οργάνων. Ε, δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε οι απαντήσεις δόθηκαν πιο πολύ γραπτός. Όλοι εκτός από το Συμβούλιο απάντησαν. Και απάντησαν με τέτοιο τρόπο που μπόρεσα να συμπεριλάβω τις απαντήσεις τους στο δικό μου σχέδιο εκθέσεως. Αν με επιτρέπετε, θα αναφερθώ καταρχάς στο Συμβούλιο. Αναφέρομαι λοιπόν στην απαλλαγή για το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο από την έποψη της Επιτροπής μας είναι συχνά το πιο προβληματικό θεσμικό όργανο και το πιο πολύ συζητημένο όργανο στο οποίο χορηγείται η απαλλαγή. Και όλοι το γνωρίζετε το θέμα αυτό. Το Συμβούλιο θα έπρεπε να είναι διαφανές θα έπρεπε να είναι πλήρως υπεύθυνο για τη χρήση των πόρων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα έπρεπε καλή την πίστη να συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία της απαλλαγής. Θα έπρεπε να διαθέτει όλα τα έγγραφα και θα έπρεπε να απαντά σε ερωτήσεις και θα έπρεπε να συμμετέχει και στις συναντήσεις με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν φορέας που ασχολείται με τον προπολογισμό παίρνει την απαλλαγή. Στην πράξη έχει αλλάξει η διαδικασία του προπολογισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ο μόνος φορέας υπεύθυνο για τον προπολογισμό ή την εκτέλεση του προπολογισμού και γι' αυτό η απαλλαγή θα πρέπει να δίδεται σε κάθε θεσμικό όργανο, σε κάθε φορέα που εκτελεί τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στείλαμε 52 ερωτήσεις στο Συμβούλιο και ακόμα απάντηση καμία. Έχω προγραμματίσει μια συνάντηση, ανεπίσημη συνάντηση, με τον πρέσβη της Ιρλανδικής Προεδρίας. Αυτό μόνο. Αλλά στόχος μας θα έπρεπε να ήταν να έχουμε επίσημες συναντήσεις με το Συμβούλιο. Και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου να συμμετέχουν στις δικέ μα συζητήσει. Αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Να έρχονται στην Επιτροπή μας. Στα πλαίσια της διαδικασίας της απαλλαγή. Προσπάθησα να κάνω κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό αποτελούσε και την βάση του θέματος που συζητάμε, αυτού που προτείνω. Από ό,τι κατάλαβα, εσείς κύριε Πρόεδρε, ως Πρόεδρος, έχετε κάποιες δυνατότητες στη διάθεσή σας. Και στο κείμενό μου άφησα τις εναλλακτικές που υπάρχουν, τις αναφέρω. Όσο δεν έχουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις μας, εγώ τι να κάνω. Δεν μπορώ να προτείνω να χορηγηθεί απαλλαγή. επομιζόμενοι τις ευθύνες. Ας αναφερθώ τώρα στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα αυτό, πρέπει να είναι ξεκάθαρα ε, ποια είναι η κατανομή των πόρων στις διάφορες κατηγορίες να μην υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά την κατανομή των πόρων στο προσωπικό, στις διάφορες βαθμίδες, στις διάφορες βαθμολογικές θέσεις. Είπαμε, το ελεγκτικό συνέδριο ενημέρωση, ενημέρωση την οικονομική και κοινωνική επίμα ενημέρωση το προσωπικό. Και αυτή η ενημέρωση για το πώς κατανέμονται τα ποσά, οι αμοιβέ στο προσωπικό αφορά και άλλα θεσμικά όργανα. Κάθε θεσμικό όργανο στην ετήσια έκθεσή του θα πρέπει να έχει έναν πίνακα. Ο πίνακα θα πρέπει να παρουσιάζει τους πόρου που δίδονται στο προσωπικό, πώ διαιρούνται οι πόροι, όχι ονομαστικά. Στατιστικά να παρουσιάσει την κατανομή των μισθών των πόρων. Ένα πίνακα που θα δείχνει πώ γίνεται η στελέχωση, ε, πώ είναι η κατανομή κατά καθήκοντα, κατά φύλλο, άντρε, γυναίκε κλπ. Η ΟΚΕ έκανε άλλα ευπρόσδεκτα βήματα προς άλλες κατευθύνσεις, προσπάθειες προσπαθεί να καλύπτει τις πραγματικές δαπάνες. Θα χρησιμοποιούνται οι νέοι κανόνες παράλληλα με το παλιό καταποκοπή σύστημα μέχρι το τέλος αυτής της θητείας. Αργότερα θα πρέπει να επιστρέφονται μόνο οι πραγματικές δαπάνες, τα πραγματικά έξοδα. Και αυτό είναι και ένα είδος απάντησης σε αυτά που ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από πέρσι οι εκπρόσωποι της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών λέγουν ότι η κοινή διοικητική συμφωνία που έχουν συνάψει έχει θετικά αποτελέσματα και για τις δύο αυτές επιτροπές και ότι είναι η πηγή μεγάλων οικονομιών. Από ό,τι φαίνεται οι αιτήσει οικονομίες εκτιμώνται στα 34,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό δεν συμπεριλαμβάνει τις οικονομίες από το μοίρασμα την κοινή χρήση αιθουσών συνεδριάσεων, κοινή χρήση εξοπλισμού στα κτίρια. Οπότε υποστηρίζω πλήρω την κοινή χρήση των χώρων και του εξοπλισμού και πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για άλλα θεσμικά όργανα. Όμως θα ήθελα να παρακαλέσω και τις δύο επιτροπές να προωθήσουν τη συνεργασία τους και να κάνουν όσες δυνατές οικονομίες υπάρχουν και όσον αφορά τη διοικητική συμφωνία θα πρέπει να βελτιωθεί ο εξορθολογισμός της χρήσης των ανθρωπίνων πόρων κυρίως των μεταφραστών. Κατά τα άλλα είμαι ικανοποιημένη με την εισαγωγή των βίντεο διασκέψεων που χρησιμοποιεί η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και προσβλέπω σε μια αξιολόγηση της μεθόδου αυτής και των οικονομιών που συνεπιφέρει. Όσον αφορά τον συνήγορο του πολίτη, να τονίσω κάτι σημαντικό και το σημείο να τονίσουμε ότι γίνεται πρόθεση του θέματος της εικόνας, διάφορα διαφημιστικά σποτάκια ε, μέσω εντύπων, μέσω διαδικτύου, προσπάθεια για ενημέρωση. Αυτός ο νέος θεσμός εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από ελάχιστους πολίτες και φορείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο διαμεσολαβητή, ο συνήγορο του πολίτη. Αυτό ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε. Ο θεσμός λοιπόν του, του εποπτικού φορέα για την προστασία των δεδομένων Πρέπει να πω ότι έγιναν διαγωνισμοί για την επιλογή προσωπικού για τις προσλήψεις, ελήφθησαν κάποια νέα μέτρα. Υπάρχει ένα νέο εσωτερικό εγχειρίδιο που δημιουργήθηκε, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια κενά όσον αφορά το προσωπικό και τις ε, προσλήψεις. Το ελεκτικό συνέδριο θα ζητά όλα τα θεσμικά όργανα να δίνουν όλα τα στοιχεία και να γίνονται έγκαιροι έλεγχοι των διαφόρων διαθεσίμων στοιχείων. Αυτό είναι κοινή πρακτική που ακολουθείται σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη, οπότε θα έπρεπε να ισχύει και για τους δικούς μας φορείς. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, παρά όλα αυτά που σας προανέφερα, παρόλα αυτά προτείνω να χορηγηθεί η απαλλαγή στα άλλα θεσμικά όργανα, στους άλλους φορείς, με την εξαίρεση του Συμβουλίου. Εξαίρεση του Συμβούλιο. Εκεί έχω και τις δύο προτάσεις. Να χορηγηθεί και να μην χορηγηθεί απαλλαγή. Έχω συμπεριλάβει και τις δύο εκδοχές. Πρότασή μου είναι όμως να αναβληθεί η απαλλαγή για το Συμβούλιο. Ε, βέβαια, είναι κάτι που μπορεί να, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης αυτό. Όμως, μέχρι τώρα το Συμβούλιο δεν απάντησε στα 52 ερωτήματα που του απευθύναμε. Και νομίζω ότι είναι δικαίωμά μας να επιμείνουμε. Και να του ζητήσουμε να μας δώσουν απάντηση από το Συμβούλιο. Θα ήθελα να διαβάσω και τα σχόλια του κυρίου Τσατνιέσκη, σχόλια που ε, αφορούν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ελεκτικό Συνέδριο. Επιτρέπετε, μπορώ. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα συνεχίσω στα αγγλικά. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης το 2011 ήταν ο πρώτος χρόνος που λειτουργήσε Δημιουργήθηκαν διάφορα τεχνικά προβλήματα που έπρεπε να ξεπεραστούν, κυρίως όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Η έκθεση συμπεριλαμβάνει διάφορα στοιχεία που μεστάλησαν γίνονται και κάποιες παρατηρήσεις από το ελεκτικό συνέδριο για μη συμμόρφωση με τους κανόνες και αφορά κάποια προβλήματα με πληρωμέ όσον αφορά το πληρωμή του προσωπικού. Υπάρχουν νομικέ αβεβαιότητε για του τους συμβασιούχους ε, ε, ορισμένου χρόνου. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση, ε, προβλήματα όσον αφορά την ανάκτηση του ΦΠΑ και τη συμμόρφωση με το δημοσιονομικό κανονισμό και μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημοσίων προμηθειών. Προτείνω ότι βασικοί δείκτες επιδόσεων θα πρέπει να καταρτιστούν για να ελέγχονται τυχόν βελτιώσεις όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού και κατά τα επόμενα χρόνια λόγω μεταφοράς μετακύλησης σε σημαντικό βαθμό διαφόρων κονδυλίων. Προτείνω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να έχει καλύτερη και πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση διότι το ποσοστό του προσωπικού που προέρχεται από τα νέα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ χαμηλό εν συγκρίση με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Εγώ θα πρότεινα να χορηγηθεί η απαλλαγή. Τώρα, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα ήθελα να πω ότι η σε λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-courier τον Νοέμβριο του 2011 συνέβαλε όσον αφορά το δικαστήριο για τη μείωση δαπανών για χαρτί κατά 25% μειώθηκε μεταξύ 2011 και 2012 οι οικονομίες είναι της τάξης των 150.000 ευρώ. Όμως οι εκκρεμούσες υποθέσεις στο δικαστήριο αυξήθηκαν από το 2010 και μετά και παρέμεινε αυτή η τάση το 2011. Άρα χρειάζεται ανθρώπινους πόρους στο δικαστήριο. Χρειάζεται βελτίωση της τελέχωσης, αύξηση τελέχωσης. Ε, χρειάζονται και άλλες θέσεις για το δικαστήριο και αυτό ε, εξετάζεται από το Συμβούλιο σαν ενδεχόμενο. Αν αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων θα μειωθεί η τάση των εκκρεμουσών υποθέσεων. Η διοικητική δομή του δικαστηρίου άλλαξε δημιουργήθηκε διεύθυνση πρωτοκόλλου και ενημέρωσης, πληροφόρησης και αναμένουμε η αιτήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 2012 να δώσει λεπτομερέστερη περιγραφή, λεπτομερή περιγραφή των ωφελιών που επέφερε η αλλαγή όσον αφορά τις επιδόσεις του δικαστηρίου. Θα ήθελα να αναφέρω ότι η απαλλαγή θα έπρεπε να χορηγηθεί. Προτείνω να χορηγηθεί. Και τέλος, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο η, ανεξ, η ανεξάρτητη μονάδα Price, ε, Water, Price, ε, Waterhouse Coopers ε, πιστεύει ότι το δημοσιονομικό δελτίο δίνει μια σωστή εικόνα της οικονομικής θέσεως του ελεκτικού συνεδρίου. Όμως χρειάζεται να σεβαστεί κάποια χρονοδιαγράμματα ακόμα και όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες χρειάζεται αυτό ειδικά να ακολουθηθεί για τις ειδικές εκθέσεις και να εθετούνται έγκαιρα πιο πολλές εκθέσεις. Όσον αφορά επικεφαλής μονάδες και διευθυντών, η ισορροπία των φύλων ε, δεν υπάρχει. Είναι πολύ... Δεν υπάρχει ισορρόπηση των δύο φύλων. Θα πρέπει να γίνεται και σωστό μοίρασμα κατά εθνικότητες περιμένουμε το 2012 να έχουμε νέα έκθεση δραστηριοτήτων όπου και την σύνοψη των βασικών πορισμάτων που απορρέουν από τον μονάδα εσωτερικού ελέγχου εκ των υστέρων εξακριβώσεων και τα αποτελέσματα των ε, αλλαγών ε, που έγιναν στον αφορά το εσωτερικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Προτείνω χορήγηση απαλλαγής στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα συνεχίσω μιλώντας τσεχικά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Γνωρίζω ότι όλα αυτά τα θέματα είναι μάλλον περίπλοκα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που μου δώσατε χρόνο για... και τη δυνατότητα να σχολιάσω την έκθεσή μου καθώς και να διαβάσω τα σχόλια του συναδέλφου του κυρίου Τσαρνιέτσκι. Βεβαίως, με τα χαράς να απαντήσω σε ερωτήσεις σας, σε σχόλιά σας. Θα ληφθούν υπόψη και θα συμπεριληφθούν και στις τροπολογίες μας. Για μία ακόμη φορά, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, που με αφήσατε να αλλάξω και τη σειρά παρουσιάσεως των εκθέσεων και της παρουσία στη σειρά αυτή που επέλεξα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. κύριε Τσέσκοβα. παρουσιάσατε και τα όσα ήθελα να πει ο κύριος ε, Τσερνέτσκι και την προηγούμενη φορά το κάνατε αυτό. Δεν ξέρω αν ο σκιώδης εισηγητής... αν οι σκιώδες είχαν τη δυνατότητα μάλλον να μιλήσουν με τον κύριο Τσερνέτσκι. Οπότε... Δεν ξέρω, ε, μιλάει ο εισηγητή με τους σκιώδες του, γιατί είναι η δεύτερη φορά που ο εισηγητή δεν είναι... Ε, παρόν στη συνεδρία της Επιτροπής. Ήθελα απλώς να το, να το θέσω αυτό. Έτσι, είμαστε όλοι βεβαίως ε, από συναδελφική αλληλεγγύη έτοιμοι να βρούμε μια ρεαλιστική λύση αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, έχω κάποιους που έχουν ζητήσει το λόγο, αλλά έχετε θέσει και ένα ερώτημα σε μένα για την ε, απαλλαγή του Συμβουλίου. Ε, το θέμα αυτό μας απασχόλησε και πέρσι. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο και τα προηγούμενα χρόνια δεν χορήγησε απαλλαγή στο Συμβούλιο. Εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής είχα την ευκαιρία και τη χρησιμοποίησα να παραστώ σε συζητήσεις με τους διαφόρους προέδρους του Συμβουλίου και να τους θέσω το θέμα αυτό και στην Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου επίσης το έθεσα ότι εμείς ως Κοινοβούλιο αυτόν τον τρόπο με τον οποίο προχωρεί το, Συμβούλιο δεν μπορούμε να τον εγκρίνουμε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Επομένως τίθεται και το ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε. Πριν ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, να θέσω ε, εγώ ένα ερώτημα. Υπάρχει κάποιος εδώ από την Ιρλανδική Προεδρία? Θα μπορούσε ίσως ο εκπρόσωπος ε, της Ιρλανδικής Προεδρίας να μιλήσει. Βεβαίως ε, μόνο να σας προσκαλέσω μπορώ, αν θέλετε μπορείτε να μιλήσετε όποια στιγμή θέλετε. Ξέρετε, το Κοινοβούλιο είναι πάντα ανοιχτό για εσάς. Απλώς ήθελα να σας καλέσω να μιλήσετε εφόσον βεβαίως η Ιρλανδική Προεδρία θέλει το λόγο έχετε πάλι τη δυνατότητα να παρέμβετε. Ωραία. Λοιπόν, να... Η κυρία Τσέσκοβα ήθελε και πάλι το λόγο για την απαλλαγή του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα, μια νέα δυνατότητα να σχολιάσω. Βεβαίως, καλέσαμε την Ιρλανδική Προεδρία ή μάλλον ήρθαμε σε επαφή με εκπροσώπους της Ιρλανδικής Προεδρίας και ζητήσαμε από την Ιρλανδική Προεδρία την ή τον εκπρόσωπο να έρθουν στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Τους είπαμε ότι θα συζητήσουμε την ε, απαλλαγή που επρόκειτο να χορηγηθεί στο Συμβούλιο και είπαμε ότι θεωρούσαμε ότι θα ήταν υπέροχο αν αυτές οι απαντήσεις είχαν απαντηθεί εγκαίρως και όπως έπρεπε, ούτω ώστε βάση ακροάσεως που διοργανώσαμε για το θέμα αυτό, μέσω ακροάσεις, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Κάποιος είχε πει νομικός ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας δεν έχει δικαίωμα για κάτι τέτοιο. Αν, θα μπορούσε κάποιος να, πει, να αμφισβητήσει κατά πόσο έχουμε την εξουσία να ζητήσουμε κάτι τέτοιο ή κατά πόσο δεν την έχουμε την έχουμε αυτή την εξουσία, προβλέπεται από τι συνθήκε. Ένα νομικό θα μπορούσε να πει ότι έχουμε το δικαίωμα, άλλο ότι δεν έχουμε. Εγώ προσωπικά επιμένω ότι έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε τι απαντήσει στι ερωτήσεις που δώσαμε επίσημα. Μέχρι τώρα όμως όπως σας είπα δεν πήραμε απάντηση. Και θα ήθελα να επαναλάβω ότι αύριο θα αυτή, θα λάβει χώρα αυτή η συνάντηση. Η Ιρλανδική Προεδρία με κάλεσε, με προσεκάλεσε να παραστώ σε αυτή τη συνεδρίαση. Πρόκειται περί ανεπίσημης συναντήσεως, όπως προανέφερα, και προσβλέπω σε κάποιο αποτέλεσμα από αυτή την συνάντηση. Προτείνω λοιπόν αυτά που σας παρουσίασα και πιστεύω ότι η άποψη της ε, Επιτροπής θα είναι ίδια όπως και με, κάποια που αυτή που ελήφθη κάποια προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ την εισηγήτρια. Υποθέτω ότι η Επιτροπή σε συμφωνία με εσά θα υποστηρίξει το έτοιμά σα, όπω και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θέλω να προκαταλάβω βέβαια στη συζήτηση. Έχω τρει ομιλητέ. Øh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δράτω με της ευκαιρίας να υποστηρίξω την ηγήτρια όσον αφορά τα θέματα του Συμβουλίου. Είναι σαφές ότι όσο δεν έχουμε απαντήσεις για τα ερωτήματα που θέτουμε δεν θα δώσουμε ε, απαλλαγή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εισηγήτρια για την αυριανή συνάντηση. Αλλά από αυτές τις άτυπες συναντήσεις τίποτα δεν βγαίνει. Ίσως να έχει κάποιες πληροφορίες η εισηγήτρια που να πιει ένα καφεδάκι μαζί κτλ. Αλλά ουσία μηδέν. Η άρνηση της χορήγησης απαλλαγής είπε ο Πρόεδρος, ε, είναι ε, συμβαδίζει με την προηγούμενη απόφασή μας. Παρ' όλα αυτά θεωρώ, όπως κάναμε και πέρσι, να δούμε τη δυνατότητα όχι απλώς αναφέροντας να θίγουμε τα ερωτήματα, αλλά να πούμε και τα ερωτήματα που είχαμε και πέρσι και, προ, και πρόπερσι. Είναι θέματα αρχής. Δεν πρέπει το Συμβούλιο να αποφύγει αυτές τις ερωτήσεις, να τις επαναλάβουμε. Να μην τις λιτώσει επειδή δεν θα έχουμε απαντήσεις. Επίσης, να πω στην εισηγητρία. Κάτι ακόμα. Ε, αρνήθηκε την αναφορά στο Gentleman's Agreement. Αυτή, αυτό που αναφέρεται στην αρχική έκθεση δεν είναι μια πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ποτέ δεν υπήρξε. 2009-10 κάναμε συζητήσεις με το Συμβούλιο, ζητήσαμε ε, να μας δώσουν κάποια έγγραφα για να αποδείξουμε την ύπαρξη αυτού του gentleman's agreement, αλλά το μόνο που είχαμε ήταν ένα έγγραφο το, στο οποίο το Συμβούλιο αναφέρεται ότι ε, μονομερός ε, δεσμεύεται σε σχέση με το Κοινοβούλιο Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η αναφορά στο Gentleman's Agreement να μην συμπεριλαμβάνεται στη φετινό μα ψήφισμα. Είναι μια συμφωνία η οποία είναι ανυπάρκτη. Ευχαριστώ. Κάλφιν. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να κάνω κάποια σχόλια για τα διάφορα θεσμικά όργανα να ξεκινήσω με τον Ευρωπαίο λεκτή Προστασία των Δεδομένων. Υποστηρίζω την πρόταση της εισηγήτριας για τον ε, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Σημειώνω την ε, σύσταση που υπάρχει στην έκθεση και την υποστηρίζω. Είναι καταρχάς αυτό το μάκρο στο οποίο τραβάνε οι έρευνες του Μεσολαβητή νομίζω ότι κρατάνε πάρα πολύ χρονικό διάστημα και καθυστερούν την όλη διαδικασία. Ε, πρέπει ίσως να, να υπάρξει καλύτερη εξήγηση για, για αυτό το θέμα. Βεβαίως δεν λέω να μην χορηγήσουμε την ε, απαλλαγή, αλλά ίσω αυτό να πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, να την ενισχύσουμε λίγο αυτή τη σύσταση. Για την Επιτροπή των Περιφερειών και την ΕΟΚΕ. Δεν έχω να πω κάτι. Για το ελεγκτικό συνέδριο, ε, συμφωνώ με τι ε, συστάσεις του εξωτερικού ελεγκτή για το ελεγκτικό συνέδριο. Ελπίζω ότι το ελεγκτικό συνέδριο θα τις εφαρμόσει τις συστάσεις του που έδωσε η Price Waterhouse Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει να συζητούμε και λόγω κάποιων πρόσφατων υποθέσεων τι θα γίνει με τις ειδικέ εκθέσεις και τι θα, πώς θα τις διαχειριστούμε και ποιος είναι ο ρόλος τελικά που έχουν να παίξουν οι ειδικέ εκθέσεις και πώς λαμβάνονται υπόψη, εάν λαμβάνονται υπόψη. Ε, νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό με, κυρίως με το ελεγκτικό συνέδριο και έχει να κάνει και με τις συζητήσεις που κάνουμε περί προϋπολογισμού. Ε, έχουμε τις προτάσεις μας, επιτάπητος, ε, πρέπει να συνεχίσουμε και ίσως να αναθεωρήσουμε την θέση του Κοινοβουλίου επ' αυτού. για το ελεγκτικό συνέδριο να ευχαριστήσω για τις γραπτές απαντήσεις που λάβαμε από την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει για το ελεγκτικό συνέδριο πάλι. Οι περισσότερες είναι απολύτως ικανοποιητικέ και συμπεριλαμβανομένες και της χρήσης ε, των ε, συστημάτων πληροφορικής και της ε, χρήσης της διαβίβασης των πληροφοριών από το από το συνέδριο, καθώς επίσης και για τους δείκτες επιδόσεων. Επίσης, ένα θέμα που θέλει περισσότερη προσοχή είναι η χρήση των γλωσσομαθών νομικών στο Λουξεμβούργο. Και η τηλεεργασία. Ε, η απάντηση του ελεκτικού συνεδρίου είναι ότι για διάφορους λόγους που κατανοώ βέβαια και τη λογική που κρύβεται πίσω από αυτή την απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που λένε είναι ότι οι γλωσσομαθείς νομικοί πρέπει να είναι είτε στο Λουξεμβούργο είτε πολύ κοντά και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν μεταφράσεις. Ίσως αυτό το θέμα να πρέπει να το ξαναδούμε. Για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Άκουσα τα σχόλια του κυρίου, που θα έκανε μάλλον ο κύριος Τσαρνέτσκι. Παρόλα αυτά, Έχω κάποια σχόλια να κάνω. Βεβαίω θα κάνω και συγκεκριμένε προτάσει ε, τι επόμενε ημέρε. Καταρχά πρέπει να πούμε σαφώ ότι ο αριθμός των θεμάτων μη ε, που, ε, των περιπτώσεων μη που εξήβρε το ελεκτικό συνέδριο ήταν πολύ μικρός και εδώ μιλούμε ούτω ή άλλω για τον πρώτο χρόνο πλήρου εργασία του προπολογισμού για την υπηρεσία εξωτερικών. Πλήρου εφαρμογή του προπολογισμού για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Τώρα, για τον αριθμό εκτέλεση. Έγιναν κάποιε σκέψει ότι δεν ήταν αρκετά υψηλό. Αυτό που βλέπουμε από τις εκθέσεις για τον ρυθμό εκτέλεσης του προπολογισμού και στα κεντρικά γραφεία και στις αντιπροσωπείες ε, είναι ότι έχει ε, αυξηθεί στο 97%. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν έχουμε να κάνουμε με την ε, ολοκλήρωση, την τελειοποίηση της τελικής εκδοχής. Επίσης υπήρξε ένα θέμα για τους βαθμούς. Κάποιοι συνάδελφοι το έθεσαν. Ε, μιλούμε για μια συγκεκριμένη περίπτωση που έχει, έχουν δοθεί κάποιες εξηγήσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει παραβίαση των κανόνων σε ό,τι αφορά την προαγωγή και τους βαθμούς στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Επίσης υπάρχει μια αναφορά στο κείμενο για την εκπαίδευση, την κατάρτιση. Αυτό πρέπει να το δούμε όμως από την πλευρά αυτού που δουλεύει εκεί. Αν εμείς αναρωτηθούμε ή ζητήσουμε από τους συναδέλφους μας, αν θεωρούν ότι θα χρειάζονταν κάποια περαιτέρω εκπαίδευση, όλοι θα απαντήσουν θετικά. Οπότε, αν πει κάποιο ότι δεν έχω τίποτα να μάθω, ε, μάλλον αυτό είναι λίγο προβληματικό, έτσι δεν είναι. Ε, Προφανώς λοιπόν το ότι το προσωπικό χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση είναι σημαντικό και δεν νομίζω ότι πρέπει να το βγάλουμε και τελείω εκτό του, του σκεπτικού μας. Επίσης για τις αντιπροσωπείες Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Ε, ο ε, επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας είναι ακριβώς ο καθήλυν αρμόδιος για διάφορες δράσεις. Επομένως, σε ένα βαθμό είναι λογικό να είναι διαφορετική εδώ η βαθμολόγηση, η βαθμολογική κλίμακα στην, στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Συμφωνώ με τα σχόλια της εισηγήτριας και του εισηγητή για την περιφερειακή ισορροπία και κυρίω ό,τι αφορά τα νεα κρατημέλη, τα νεοτερα κρατημέλη. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δούμε και το πώς δημιουργήθηκε αυτή η υπηρεσία. Κυρίως στελεχώθηκε από ε, προσωπικό που ήδη εργάζεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σιγά σιγά το ποσοστό ε, από τις εθνικές, ευρωπαϊκές, από αυξήθηκε. Είμαστε περίπου στο 1 τρίτο του προσωπικού Πρέπει όμως να δούμε και την τάση η οποία υπάρχει και είναι αυξητική. Και αυτό βεβαίω πρέπει να το ενθαρρύνουμε. Τέλος, για το Συμβούλιο. Δεν θα μπορούσα να πω τίποτα διαφορετικό από όλα όσα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το Συμβούλιο πρέπει να παρουσιάσει τις πληροφορίες που το έχουμε ζητήσει. Πρέπει να μα πει τι πιστεύει για την απαλλαγή και για το ρόλο του Κοινοβουλίου. Δεν γίνεται να μην απαντά. όχι μόνο ω ε, ευρωβουλευτέ, αλλά και ω πολίτες περιμένουμε απαντήσει από το Συμβούλιο. Οπότε, Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν να ξαναθέσουμε το θέμα αυτό είτε σε κάποιο θεσμικό όργανο, είτε στο ελεκτικό συνέδριο που μπορεί τελικά να μας δώσει μια απάντηση στο τι τελικά ρόλο παίζει το Κοινοβούλιο στην όλη διαδικασία ε, απαλλαγή. Δεν αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα όταν θέτουμε συνέχεια ερωτήσει στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο απλώ αρνείται να απαντήσει. Οπότε είμαι υπέρ τη ε, πρόταση τη συγκίτρια να αναβάλουμε την απαλλαγή προ το παρόν και θα ήθελα να δούμε πώ θα λύσουμε το θέμα αυτό. Αν δεν μπορούμε να το λύσουμε μεταξύ μα, δηλαδή μεταξύ των δύο θεσμικών ε, οργάνων, α βρούμε έναν διαιτητή που μόνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να είναι για να μας πει ποιος είναι ο ρόλος του καθενός στην όλη διαδικασία απαλλαγής. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Επόμενος, ο κύριος Ροντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ την εισηγήτρια για το δύσκολο έργο για να συντάξει αυτή την έκθεση. Μεγάλη, πολλή δουλειά για την απαλλαγή στο Συμβούλιο και, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αν κατάλαβα καλά, προσανατολιζόμαστε σε μια αναβολή της απαλλαγής στο Συμβούλιο και θα δώσουμε απαλλαγή στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τεχνικά, ποιος είναι ο λόγος, ποιο, ε, τα επιχειρήματα και η αιτιολογία να μην δοθεί απαλλαγή στο Συμβούλιο της Ευρώπης ή και να δοθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ποια είναι τα θέματα. Απάντησε το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 52 ερωτήματα και δεν το έπραξε το Συμβούλιο. Τι γίνεται ακριβώς. Εγώ είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι η, η, αρχή που ελέγχει όλες τις, ε, όλα τα όργανα είναι το ελεκτικό συνέδριο και εγώ ενδιαφέρομαι να ξέρω τη γνώμη του ελεκτικού συνεδρίου για να ξέρω πώς ακριβώς αυτό θεωρεί το θέμα διότι είναι το, το πλεισμένο μας χέρι θα έλεγα το ελεκτικό συνέδριο. Όταν βλέπω την έκθεσή του δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω για τα διάφορα θέματα υπάρχει μια παρατήρηση κάτι για ε, κάποια αγορά ε, υλικού, αλλά δεν, γενικά δεν βλέπω τίποτα, τίποτα, τίποτα το ιδιαίτερο. Ε, χρόνια γίνεται τώρα αυτή η συζήτηση. Αν, ε, αν κάνουμε μια αναβολή στην απαλλαγή που θα οδηγήσει σε άρνηση τον Οκτώβριο, δηλαδή ποιε θα είναι οι επιπτώσει, οι κυρώσει στο προσωπικό. Θα ήθελα μια ανταλλαγή απόψε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια σε αυτή την κατάσταση. Θέτω λοιπόν το ερώτημα στη συζήτρια μας. Γιατί ε, δεν δίνει, αρνείται την απαλλαγή στο Συμβούλιο και όχι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τι ακριβώς γίνεται. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ αντικαθιστώ προς τον παρόν τον ε, πρόεδρο. Ο κύριος Γκάιερ έχει πρώτα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα για, τον, ε, για το θέμα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Συμμερίζομαι τις ε, προτάσεις της εισηγήτριας απόλυτα και ο συνάδελφος Κάλφιν είπε ακριβώς ε, αυτά εξ ονόματος της ομάδας μας αλλά θέλω δύο πράγματα να θέσω προς συζήτηση. Δεν πρέπει ή ίσως να μην μπορούμε κιόλας να τα ολοκληρώσουμε σήμερα αλλά ίσως θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν λίγο παρακάτω. Λοιπόν, κάναμε για αυτό το θέμα μία ακρόαση. Και, και οι δύο προσκεκλημένοι, οι εμπειρογνώμονες, ε, ήτανε, ε, δεν συμφωνούσαν για το τι γίνεται με τις συμβάσεις και για την, απο, για την απόφαση απαλλαγής του Συμβουλίου. Σε ένα πράγμα όμως συμφωνούσανε. Στο ερώτημα του αν έχει το, ε, το Κοινοβούλιο το, δικαίω, το δικαίωμα να λάβει τις πληροφορίες αυτές από όλη τη διαδικασία. Εκεί υπήρξε απόλυτη συμφωνία των προσκεκλημένων. Στο παρελθόν, για το θέμα της απαλλαγής του Συμβουλίου, ε, για το σε ό,τι αφορά το πόσο ισχυρό είναι το δικό μα όπλο. Έκανα κάποιε παρατηρήσεις, το είπε και ο κύριος ε, Ροντή. Η δική μου ομάδα βέβαια μέχρι στιγμής ήταν απομονωμένη για το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι για το σημείο αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι ότι το Συμβούλιο αυτή την διαφάνεια που του ζητούμε πρέπει να την τηρήσει. Αν τώρα υπάρχει η συμφωνία από του εμπειρογνώμονε ότι εμεί έχουμε το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να έχουμε συγκεκριμένα έγγραφα μπροστά μα, τότε εγώ θα ήθελα να το εξετάσουμε αν για αυτό το σημείο μπορεί να παρέμβει το δικαστήριο. Για το θέμα δηλαδή της προσβασιμότητας των εγγράφων. Δεν μιλώ για την απαλλαγή αυτή καθ' αυτή. Ε, εκεί ίσω να υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που ουσιαστικά θα μας βάλει σε μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι θα μας προχωρήσει. Αλλά σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα των εγγράφων θα πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Και ίσως ο πολύ ε, συμπαθής εκπρόσωπος της Ιρλανδικής Προεδρίας να το θέσει αυτό προς συζήτηση. Το, το Κοινοβούλιο έχει πάρα πολλά θέματα να συζητήσει με το Συμβούλιο και για θέματα ε, καλύτερων δαπανών, διαφάνεια, προπολογισμού. Εμεί εδώ ω ως, ως Κοινοβούλιο ε, έχουμε μπει σε μια διαδικασία με το, με το Ελεκτικό Συνέδριο και το Συμβούλιο, εάν εμεί έχουμε το, το δικαίωμα να λάβουμε έγγραφα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα που θέλω να, να θίξω. Έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Έχω κάποια προβλήματα όταν η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για ένα τέτοιο ε, θεσμικό έργανο που είναι υπεύθυνο για όλα όσα έχουν να κάνουν με χρήματα και που μιλάμε και για μισθούς δηλαδή ε, είμαι λίγο διστακτικός αν για ένα τέτοιο θεσμικό όργανο μπορούμε να συμπεριλάβουμε ένα σημείο ως απλή τροπολογία. Ανεξάρτητα από το θέμα, το ερώτημα μάλλον που θέλω να θέσω. Στα ΜΜΕ ε, συχνά ακούμε ε, ότι το ε, ελεκτικό συνέδριο έχει ένα γραφείο του πρώην βουλγαρικού μέλους του ελεκτικού συνεδρίου το οποίο είχε μπλακεί σε πολλές παράνομες δραστηριότητε. Το κολέγιο του ελεκτικού συνεδρίου αποφάσισε και έτσι κατάλαβα εγώ ότι δεν θα πάνε αυτές οι υποθέσεις στο δικαστήριο. Το ερώτημα τώρα αν οι υπάλληλοι ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων μπορούν να, ε, κάνουν, να έχουν μια τέτοια δραστηριότητα, είτε είναι μέλη του, του ελεκτικού συνεδρίου, είτε είναι άλλα υψηλά μέλη της, ε, του, των θεσμικών οργάνων. Αν μπορούν να έχουν μια τέτοια συμπεριφορά, ε, δεν ξέρω, σίγουρα αυτό δεν ανήκει στο θέμα της απαλλαγής, αλλά το θέμα του πώς διαχειρίζεται αυτές τις υποθέσεις που το αφορούν το ελεκτικό συνέδριο και αν αυτό έχει να κάνει με το ε, αν μπορούμε να υποβάλουμε κάποιο αίτημα για την ε, πρόθεση αυτής της ε, υπόθεσης και προς το ελεγκτικό συνέδριο, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Πρέπει να και οι πολίτες να ξέρουν ότι υπάρχουν συνέπειες όταν υπάρχουν παράνομες συμπεριφορές και ότι δεν υπάρχουν ε, ε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο Γενικό Γραμματέα είναι εδώ, οπότε θα ήθελα παρακαλώ, αν μπορεί, να μα απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Γκάιερ. Ο κύριος Κυλακάκης έχει το λόγο. Ε, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προσπάθειες που κατέβαλε Όσον αφορά το Συμβούλιο δεν έχω τίποτα περισσότερο να πω. Συμφωνώ με τους προλαλήσατες, δεν μπορούμε να χορηγήσουμε όσοι έχουν τα πράγματα την απαλλαγή, θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, το συζητήσαμε αυτό λεπτομερώς σε προηγούμενες περιστάσεις. Θα ήθελα να προσθέσω απλώς ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, έχει μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου που συντάσσει εκθέσεις σχετικά με τα όσα γίνονται και μας ενδιαφέρουν αυτές οι εκθέσεις. Ενδιαφέρουν το ελεκτικό συνέδριο και θα πρέπει να εξετάσουμε λεπτομεράστερα τα θέματα διότι είναι μια αρχή αυτή, καινούργια αρχή Ποιο τμήμα, ποιο κομμάτι των εκθέσεων αυτών μπορούμε να δούμε εμείς και το ελεκτικό συνέδριο. Για το δικαστήριο το ευρωπαϊκό να πω ότι βλέπουμε σημαντική αύξηση αναφέρει ο συγκεκριτής σημαντική αύξηση εκκρεμωδικιών. Ε, ε, είναι πολύ σημαντικό θέμα διότι η αύξηση των εκκρεμωτήτων, εκκρεμών υποθέσεων σημαίνει λιγότερη ασφάλεια δικαίου ε, στην Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να εξεταστεί διότι είναι σημαντικό θέμα επηρεάζει τις οικονομίες όλων διότι πολλά εξαρτώνται από τις αποφάσεις του δικαστηρίου και ίσως κάτι πρέπει να κάνουμε ή να το συζητήσουμε λεπτομερέστερα τουλάχιστον αυτό Όσον αφορά το ελεγκτικό συνέδριο, θα ήθελα να πω ότι αυξάνεται δυσαρέσκεια των εξωτερικών ε, όσον αφορά τους εξωτερικούς ελεγκτές που χρησιμοποιεί το ελεγκτικό συνέδριο. Θα ήθελα λεπτομέρειες από πλευράς του εισηγητή. Γιατί υπάρχει αυτή η αύξηση δυσαρέσκειας Αυτό πρέπει να εξεταστεί. Για την ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή χρειάζεται λεπτομερέστερη ανάλυση και κάτι άλλο. Προσωπικό το οποίο που έχει προσληφθεί από την Επίτροπη και κατά πόσο υπάρχουν προβλήματα στην όλη διαδικασία. Και αυτό πρέπει να εξεταστεί ενδελεχέστερα. Και τέλος, για τον Ευρωπαίο, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, το συνήγορο του πολίτη, συμφωνώ με τον συνάδελφο, πράγματι πρέπει να εξετάσουμε γιατί χρειάζεται περισσότερο χρόνο όσον αφορά τις έρευνες που διεξάγει ο συνήγορος του πολίτη. Δεν αρκούν τα χρήματα, είναι μικρό ο υπολογισμός, υπάρχει πρόβλημα με τα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη λειτουργία του θεσμού. Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί λεπτομερέστερα. Εν γέννη, συμφωνώ με τις συστάσεις του εισηγητού και σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Τάμπας Ντόιτς, επόμενος. Eh, ευχαριστώ. Καταρχάς, να πω ότι ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. Θα μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Ρούμπιχ στην αρχή της ε, συνεδρίασης. Είναι όντως πολύ περίπλοκο το θέμα και θα πρέπει όντως να εκφραζόμαστε πολύ συγκεκριμένα και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι ε, απολύτως ακριβής. Δεν θα σχολιάσω αυτά για τα οποία συμφωνώ. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις για τροπολογίες, ε, τις οποίες βεβαίως θα υποβάλλω και γι' αυτό δεν θέλω να, τις, ε, να τα σχολιάσω όλα αυτά, μια που έχουμε και πολύ λίγο χρόνο, αλλά δεν θέλω και να καθυστερήσω τη διαδικασία με τα, επαναλαμβάνοντας τα σχόλια των ε, όσων πήραν το λόγο. Τέσσερα πράγματα θέλω να πω μονάχα και θα ξεκινήσω με την ε, απαλλαγή του Συμβουλίου. Καταρχάς διαπιστώνω ότι δεν είναι σοβαρή η θέση του Συμβουλίου. Μπορεί να εκφράζομαι λίγο απότομα, αλλά νομίζω ότι περιγράφει ακριβώς το, την συμπεριφορά του Συμβουλίου εδώ και καιρό. Και πρέπει να πω ότι εδώ είμαι στο, εγώ είμαι στο Κοινοβούλιο εδώ και 3,5 χρόνια. Δεν έχω την τεράστια εμπειρία, αλλά παρόλα αυτά αμφιβάλλω για το ότι και από πολιτική και από νομική πλευρά μιλούμε για την θέση εδώ του ε, Συμβουλίου. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ο κύριος Ρομπάι ως μόνιμος πρόεδρος. Α, παλιά δεν υπήρχε γιατί δεν υπήρχε η θέση. Τότε υπήρχε η θέση του Συμβουλίου και ένας πρόεδρος του Συμβουλίου ε, άλλαζε μετά το ένας μετά τον άλλον κάθε έξι μήνες. Όπως ξέραμε αυτό παραμένει το ίδιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους διαφόρους εκπροσώπους του Συμβουλίου, στην Ολομέλεια, αλλά και εδώ, λένε ότι θέλουν να αλλάξει το θέμα αυτό, αλλά παρόλα αυτά δεν κάνουν τίποτα για να αλλάξει. Ε, Και γι' αυτό φοβόμασταν κάποια στιγμή τι ακριβώς θα αρχίσουν να σκέφτονται οι ε, ψηφοφόροι, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αλλά εδώ μιλούμε για την γραφειοκρατία του Συμβουλίου, η οποία έχει μια θέση και η θέση αυτή εκφράζεται ακριβώς μέσω του μόνιμου Προέδρου του Συμβουλίου, είτε του ε, εκ ε, είτε της χώρας που αναλαμβάνει την εκπεριτροπής προεδρία. Είναι νομίζω γραφειοκρατική η θέση αυτή. Ε, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που περιμένουμε ή που θα σκεφτόμασταν ότι πρέπει να είναι η θέση ενός θεσμικού οργάνου. Βεβαίως όλοι αυτοί οι γραφειοκράτες στο Συμβούλιο είναι πάρα πολύ καλοί υπάλληλοι, μορφωμένοι, αλλά το κοινοβούλιο ε, νομίζω ότι δεν του δίδεται από το Συμβούλιο τουλάχιστον ε, η σημασία που πρέπει. Ε, ίσως σε έναν υπηαγωγείο τα παιδιά να μπορούσαν να λύσουν πιο εύκολα το πρόβλημά τους από ότι μπορούμε εμείς να λύσουμε το πρόβλημά μας με το Συμβούλιο. Τώρα, για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Για το θέμα των ακινήτων, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και θα πρέπει να υποβληθούν κάποιες τροπολογίες σε σχέση με το σχέδιο έκθεσης. Καταρχάς, πιστεύω ότι η κυρία Άστον ε, έχει δώσει, την, ε, έχει αναφέρει μάλλον ότι αυτή ότι όντω θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση για τα, για τα ακίνητα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Καλό λοιπόν θα ήταν αν μπορούσε να διευκρινιστεί το θέμα αυτό. Ξέρουμε πώς έχουν αυτές οι συμβάσεις. Δεύτερον, νομίζω ότι είναι τελείως απαράδεκτο η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων να κάνει εσωτερικό έλεγχο και μετά να κάνει μια αξιολόγηση για τη διαχείριση των εκινητων Και μετά να λένε ότι εμείς δεν θα έχουμε καμία άποψη, καμία, ε, ούτε καν θα δούμε αυτό το υλικό. Νομίζω ότι κατά αυτή η προσέγγιση. Ε, εφόσον μιλούμε για την ε, διαχείριση των ακινήτων και μιλούμε και για, την, για τον έλεγχο ακριβώς αυτής της διαχείρισης, μία ε, βιβλιογραφία θα μας βοηθούσε. Θα βοηθούσε να έχουμε κι εμείς μία τεκμηρίωση στα χέρια μας. Γι' αυτό θα πρέπει κι εμείς να έχουμε άποψη για το θέμα αυτό. Και άλλη μία παρατήρηση Νομίζω ότι δεν εκφράζεται σωστά στην έκθεση το, το θέμα των ε, μισθών, ε, των ε, υπαλλήλων που πρέπει να ισοσταθμιστεί με τον μισθό των υπαλλήλων του ΝΑΤΟ. Ίσως κάποια στιγμή η χρονική να είναι καλή, αλλά η σημερινή χρονική στιγμή δεν είναι η κατάλληλη. Νομίζω ότι το κείμενο που έχουμε λάβει από το ελεγκτικό συνέδριο δείχνει ότι υπάρχουν πραγματικά τεράστιες ανισορροπίες και σε ό,τι αφορά την εθνικότητα των μελών του, Ελεκτικού Συνεδρίου και αυτό πρέπει να λυθεί. Και θα επανέλθω σε αυτό που είπε ο κύριος Κυλακάκης για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, είναι όντως ε, το θέμα αυτό αρκετά κανθόδες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το δικαστήριο πρέπει να παρέμβει αποτελεσματικά. Και μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο αν δούμε ότι όντω χρειάζονται περισσότεροι υπάλληλοι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να κάνει τη δουλειά του, ε, τότε ίσως να είναι σημαντικό να δώσουμε αυτά τα έξτρα κονδύλια. Έστω και αν δεν μπορούμε βραχυπρόθεσμα να εξοικονομήσουμε ε, κονδύλια. Συμφωνώ λοιπόν με τον ε, Ευρωβουλευτή ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Ντόιτς. Η κυρία Γκρέσλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Για το ε, ελεκτικό συνέδριο και για τις ε, υποθέσεις αυτές που ακούσαμε, νομίζω ότι θα πάνε στο δικαστήριο. Οπότε το θέμα των ε, υπαλλήλων του, ε, του Ανοιχτικού Συνεδρίου νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους για το τι θα γίνει. Τώρα, ο συνάδελφος Σοντή πάντα έχει μια δική του ιδιαίτερη άποψη εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, όλοι νομίζω ότι συμφωνούμε τα μας ότι δεν μπορούμε να δώσουμε απαλλαγή στο Συμβούλιο που δεν μας ε, ε, δίνει καμία, κανένα λογαριασμό για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, προφανώς αυτό είναι εκ των ανουκάνευ. Ούτως ή άλλως αυτό πρέπει να ε, συνδεθεί και, με, τον, ε, και τη συζήτηση, με τη συζήτηση για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να τα ξεκαθαρίσει τα θέματα αυτά. Αν δεν θέλει να δώσει παραπάνω λεφτά, τουλάχιστον θα πρέπει να ε, ξεκαθαρίσει τα όσα έχει διαχειριστεί μέχρι τώρα. Τώρα, για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων η κυρία Τσέσκοβα δεν φταίει, αλλά απογοητεύτηκα λίγο γιατί είναι η πρώτη απαλλαγή τη Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και ήθελα λίγο περισσότερη τάξη στην έκθεση. Θα μπορούσαμε α πούμε, να μιλήσουμε ξεχωριστά για τα κεντρικά γραφεία και ξεχωριστά για τι αντιπροσωπείες και εκεί θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε ε, τα, τις ροές, τις οικονομικές, το προσωπικό. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία ναι, μεν είναι θετικά, είναι ενδιαφέροντα. Το λυπηρό είναι ότι είναι όλα λίγο ανάμεικτα. Ε, κρίμα. Ίσως την επόμενη φορά να μπορούσαμε να, να, παρέμβουν λίγο πιο νωρίς. Ε, και έρχομαι από μια συζήτηση ακριβώς για τον, ε, από μια, που έγινε στην, για, ακριβώς για το θέμα του προπλογισμού και η εσωτερική αναθεώρηση, η ιστορική αυτή έκθεση έχει να κάνει με την αλλαγή του προϋπολογισμού και αυτό ήταν η προϋπόθεση για να, να... να αποσυνδεθεί από την Κομισιόν η ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων, ότι δηλαδή θα είναι καθαρή προ τα οικονομικά της απέναντί μα. Η υπεύθυνη, η επικεφαλής της αντιπροσωπείας έχει, το, έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται κονδύλια τα οποία βεβαίως κατανέμονται μέσα στην, στην υπηρεσία. Έχουμε 36 ουσιαστικά 36 αντιπροσωπείες που έχουν ένα άτομο. Δηλαδή μόνος του ο πρεσβευτής είναι μόνος, αποτελεί μόνος του την αντιπροσωπεία. Λοιπόν, ε, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση για αποτελεσματικότητα είτε δεν θα χρησιμοποιούμε πια αυτές τις ε, ε, αντιπροσωπείε, είτε θα τι εμπλουτίσουμε, θα τι ε, στελεχώσουμε περισσότερο δυναμικό, με περισσότερο προσωπικό για να μπορεί κανεί να κάνει τη δουλειά του. Γιατί δεν μιλούμε μόνο για χρήματα της Κομισιόν, μιλούμε για την, τη δική τους οικονομική διαχείριση. Η Κομισιόν ουσιαστικά ρυθμίζει την οικονομική διαχείριση της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό αν παρεκκλίνουμε από το, χρέο χρέος που έχει το κάθε θεσμικό όργανο να δίνει λογαριασμό για τα κονδύλια του, εμείς πώς θα μπορέσουμε να, να θέσουμε επί των, ε, ε, ενώπιον ευθυνών την, Κομισιόν που έχει δώσει τα διάφορα κονδύλια στι διάφορες υπηρεσίε. Οπότε αυτό είναι πολύ ανησυχητικό γιατί μιλούμε για ένα ε, δικαίωμα εδώ, που ισχύει εδώ και 50 χρόνια το δικαίωμα της λογοδοσίας. Και Νομίζω ότι αυτά τα θέματα είναι ιδιαίτερο σημαντικά ε, και συνήθως τα διαχειρίζονται άνθρωποι που δεν έχουν έτσι πολύ καλή κατανόηση των μεγάλων, ε, της μεγάλης εικόνας του γενικού οράματος. Για τα όσα είπε ο συνάδελφος Κάλφιν. Μίλησε για την ε, περαιτέρω εκπαίδευση, την κατάρτιση. Ο συνάδελφος Τσαρνέτσκι ε, δικαίω νομίζω διαπιστώνει ότι για πρώτη φορά έχουμε εκθέσεις από όλες τις αντιπροσωπείε. Λάβαμε 136 ε, εκθέσει αντιπροσωπιών και πάνω από τις μισές παρατηρούν ότι οι συνεργάτες δεν έχουν τα προσόντα για τα καθήκοντα τα οποία έχουν αναλάβει και γι' αυτό χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική διαπίστωση. Δεν λέμε ότι όλου θέλουμε να του εκπαιδεύσουμε περαιτέρω. Όχι, αλλά αυτό έχει να κάνει με το πώ διαχειριζόμαστε, μάλλον πώ αυτή η υπηρεσία κάνει τη δουλειά τη. Ποια είναι τα μέσα που έχει για να μπορεί να κάνει τη δουλειά τη. Γι' αυτό θέλω να ζητήσω αυτό το σημείο να παραμείνει στο κείμενο. Για πρώτη φορά έχουμε λάβει εκθέσει από τι εθνικέ αντιπροσωπείε. Θα ήθελα να, να τύχουν μεγαλύτερη ε, προσοχής. Είναι σημαντικά έγγραφα. Ναι, είναι σημαντική η δουλειά που έχει γίνει. Ε, πρέπει να περάσει και σε φόρματα Excel για να τη διαβάσουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικά αυτά που περιλαμβάνουν και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα. Επίση, ο συνάδελφο Κάλφιν είπε ότι ο αριθμό των ε, συνεργατών δεν φτάνει, από τα κρατημέλη δηλαδή. Ένα τρίτο είπε των ε, υψηλών θέσεων πάει σε εκπροσώπους κρατών μελών. Και από αυτό το 1 τρίτο έχουμε ε, ουσιαστικά δεν έχουμε ούτε, ούτε διαγωνισμούς, ούτε τίποτα. Κατελείεται δηλαδή και, το, και ο, δικό, ο ευρωπαϊκός κανονισμός ό,τι αφορά την στελέχωση θέσεων. Ακριβώς λοιπόν αυτό το, τον, το ότι ο, ο, θα, θα προσληφθεί αυτός που έχει τη μεγαλύτερη πίεση ή ο φίλος του φίλου, το έχουμε διαπιστώσει. Γι' αυτό θα ήθελα αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ θέλω να υπερασπιστώ τον ιστορικό κανονισμό, γιατί ακριβώς σε αυτό το σημείο υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη και τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλους. Γι' αυτό, αυτό το σημείο, ε, είναι, σε αυτό το σημείο είμαι αντίθετη με τον κύριο Κάλφιν. «39% των ε, θέσεων πάνε περίπου στις, ε, μάλλον ε, ε, ένα τρίτο είναι στις, που πάει στις θέσεις από εκπροσώπους κρατών μελών και όχι το 39%. Και επίσης, ήμουνα στην διάσκεψη των Προέδρων και άκουσα διάφορες ωραίες ομιλίες για την Ευρώπη για το πόσο Ευρωπαίοι είμαστε σε μια εξωτερική υπηρεσία δράσεων, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική ερώτηση. θα αφήσουμε τα κράτη-μέλη να, πάρουν, να πάρει ο καθένα σε τη θέση που θέλει ή θα θέσουμε ευρωπαϊκά κριτήρια, κοινά κριτήρια για όλου τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται. Εγώ προφανώ είμαι υπέρ τη δεύτερη επιλογή. Γι' αυτό συμφωνώ με τον συνάδελφο Τάμα Στόιτ. Ε, θα κάνουμε κάποιε τροπολογίε έτσι ώστε να εμπλουτιστεί το κείμενο, το οποίο όμως ούτως ή άλλως είναι καλό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Γκρέσλε. Κλείνοντας, η κυρία κυρια γκρεσλε κλείνοντα η κυρια ανδρεασεν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εστιαστώ στην υπηρεσία εξωτερική δράση και στο Συμβούλιο. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων, μερικά σχόλια ακούστηκαν με τα οποία συμφωνώ, αλλά ανησυχώ βασικά για το εξή. Θεωρείται ότι ο αριθμό των σφαλμάτων και ατασταλιών που βρέθηκαν φαίνεται να είναι μικρός και ότι είναι ασήμαντα τα σφάλματα σε βαθμό που θέλουμε να τους δώσουμε απαλλαγή. Λυπάμαι. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι ένας νέος θεσμός και πρέπει να είμαστε αυστηρότεροι ε, απαιτώντας αποτελεσματικούς ελέγχους ούτως ώστε να αποφύγουμε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με άλλους φορείς κατά τα περασμένα χρόνια αισθάνομαι ότι είμαι σε δύσκολη θέση. Ξεκινά ένας νέος θεσμό, ένα νέο όργανο και έχουμε προβλήματα με τις προμήθειε και τις προσλήψεις. Έχουμε προβλήματα με τις αμοιβέ των ε, μελών του προσωπικού. Και παρόλο που η στελέχωση είναι αρκετά μικρή, έχουμε μεγάλα προβλήματα. Έχω μεγάλα προβλήματα μαθαίνοντας ότι ότι έχουμε μεγάλη μεταφορά μετακύληση κονδυλίων. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε σωστή διαδικασία διαθέσεως κονδυλίων προς την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και είναι ένα νέο ε, όργανο θα έπρεπε να μετακινηθούμε από τις ατασταλίες των διαδικασιών και να μετακινηθούμε και να κρίνουμε την απόδοση που έχουν τα διάφορα, διάφοροι οργανισμοί. Και αν κάπου έπρεπε να εστιαστούμε είναι στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Διότι στο κάτω-κάτω έχει αυξανόμενη ε, επίδραση όσον αφορά τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κατά την άποψή μου, ε, δεν θα έλεγα να δώσουμε απαλλαγή στην υπηρεσία, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα του ζητούσα, θα ζητούσα από τη Βαρόνη Άστον ένα οργανόγραμμα, ένα σχεδιασμό. Ε, πώς θα χειριστεί την ε, διοίκηση αυτού του φορέα τον επόμενο χρόνο και πώς μπορεί να είναι βέβαιοι ότι οι ελλείψεις που διαπιστώσαμε κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και τα κενά δεν θα επαναληφθούν. Όσον αφορά το Συμβούλιο, ε, συζητούσαμε την απαλλαγή προς το Συμβούλιο επί μακρόν. Όσο είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ίσως και πριν από αυτό, το συζητούσαμε. Και νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια πρακτική λύση. Πρώτα απ' όλα, δεν είδα στην έκθεση του ενεκτικού συνεδρίου το ίδιο επίπεδο επικρίσεων κατά του Συμβουλίου όπως για άλλα θεσμικά όργανα. Άρα θα πρέπει να είμαστε προβληματισμένοι όσον αφορά τη δίκαιη αντιμετώπιση. Γιατί επικρίνουμε ε, με δρυμύτητα το Συμβούλιο επειδή δεν μας απαντούν, δεν απάντησαν στα 52 μας ερωτήματα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί διότι είδα κενά σε άλλα θεσμικά όργανα τα οποία είναι λιγότερο σημαντικά από αυτά που, από το Συμβούλιο. Και το θέμα της αμοιβαιότητα. Δεν ξέρω, συζητήσαμε με το Συμβούλιο. Εμείς μπορούμε να ανοίξουμε τα βιβλία του Κοινοβουλίου. Αν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό, μήπως θα ανταποκρινόταν καλύτερα το Συμβούλιο από ό,τι σήμερα διότι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν απαντούν ή δεν δίνουν ε, πληροφορίες είναι ότι το Κοινοβούλιο δεν ανοίγει τα βιβλία του στο Συμβούλιο. Γιατί να μην ανοίγουμε εμείς τα δικά μας βιβλία προς το Συμβούλιο. Ρωτάω. You know, back to the Τώρα να μπούμε στα, στις πρακτικές λεπτομέρειες. Μέχρι τώρα ήδη ε, δεν έχουμε χορηγήσει την απαλλαγή και δεν συνέβη τίποτα με το Συμβούλιο. Τι περιμένουμε τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, τι περιμένουμε. Μπορούμε να μην χορηγήσουμε την απαλλαγή για ένα, δύο, τρία χρόνια και δεν τους νοιάζει καθόλου. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο και τι τους νοιάζει. Μειώσανε τον προπολογισμό για τα επόμενα αυτά χρόνια, δεν τους νοιάζει. Λοιπόν, εάν σταματήσουμε τη χρηματοδότησή τους, γιατί οι δικές τους διοικητικές δαπάνες μέχρι ότου ανοίξουν τα βιβλία τους, γιατί δεν αποφασίζουμε κάτι τέτοιο, να παρακρατήσουμε τους πόρους τους, τους σχετικούς με τις δικές, δικές τους διοικητικές δαπάνες, τις δικές τους επιχειρησιακές δαπάνες. Γιατί να μην εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας, πώς να το πω, τέτοιας Ευχαριστώ κύριε Ανδρέασεν. Ο κύριος Σοντή έχει ξαναζητήσει το λόγο. Να σας πω ότι αυτό το δύσκολο ερώτημα σίγουρα δεν θα το ολοκληρώσουμε σήμερα. Ε, Ήδη είχαμε, έχουμε ακολουθήσει το δρόμο αυτό εδώ και πολλά χρόνια και η θέση της, ε, του Κοινοβουλίου μέσω της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού είναι σαφής. Βεβαίως είμαστε υπέρ της διαφάνειας. Το Κοινοβούλιο είναι ουσιοδός διαφανέστερο. Έχουμε θέσει λοιπόν διάφορα ερωτήματα, έχουμε απαντήσει, αλλά μπορούμε να το δούμε το θέμα από διάφορες οπτικές γωνίες. Η κυρία Τσέσκοβα μίλησε για την νομική πτυχή του θέματος. Έχουμε και ένα εργαστήριο του Κοινοβουλίου όπου τα νομικά θέματα ακριβώς ετέθησαν και υπήρξαν και διάφορες απόψεις εκεί για το κατά πόσο το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να απαλλάξει το Συμβούλιο αλλά σε ένα νομικό θέμα όλοι οι νομικοί που είχαμε καλέσει ήταν τη ίδια άποψη. Ότι δηλαδή το Κοινοβούλιο έχει το αναφέρετο δικαίωμα ε, θέματα, ερωτήματα που θέτουμε να, απαντούν, να απαντώνται. Οπότε τίθεται το ερώτημα, εάν ε, δεν καταλήξουμε σε μια λύση, αυτό το, πράγμα, αυτό το θέμα δεν πρέπει να ξεκαθαριστεί από το, από το δικαστήριο, όπως είπε και ο κύριος Κάλφιν αν δεν το λύσουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, περνάει ο χρόνος και επειδή έχουμε και άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη για σήμερα, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντί και μετά στην εισηγήτρια. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να εφαρμόσουμε το δίκαιο, συμφωνώ, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό. Σε όλε τι δημοκρατίε υπάρχει ένα κοινοβούλιο το οποίο ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Ζήτησα ε, να υπάρχει παρουσία του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Ε, να καλέσουμε ίσω τον κύριο Φαναρπόη να μα πει ποια είναι η άποψή του για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ίσως να καλέσουμε αυτούς που ήταν στην Προεδρία το 2011. Η η Ιρλανδική Προεδρία ίσως ε, να μας πει κάτι. Κάποιοι αρμόδιοι, κάποιοι υπάλληλοι να μας δώσουν να καταλάβουμε πώς έχουν τα θέματα και πώς μπορούμε να ασκήσουμε έλεγχο στο, στην εκτελεστική θα λέγαμε εξουσία. Ευχαριστώ. Προς ενημέρωση. Ω πρόεδρο τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, βεβαίω έχω επαφέ με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Ρομπάη. Έχουμε συζητήσει εντατικά για το θέμα του προπολογισμού και της μεσοπρόθεσμου, του μεσοπρόθεσμου πλαισίου και του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού. Αλλά βεβαίω μου είπε ότι ο αυτός είναι ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όχι ο πρόεδρο του Συμβουλίου. Οπότε δεν είναι υπεύθυνο για την απαλλαγή. Η υπεύθυνη είναι η Ιρλανδική Προεδρία ή η επόμενη Προεδρία, η εκπεριτροπή Προεδρία. Οπότε αύριο ε, θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό, όχι για την απαλλαγή, αλλά για άλλα θέματα. Ε, εντάξει, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το θέσουμε. Εγώ έχω έρθει σε επαφή και με τον ε, Υπουργό Χέι. ε, και ακριβώς του έθεσα το θέμα αυτό. Ε, το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι ο, η συγκήτρια αλλά και η κυρία Τσέσκοβα αλλά και η Ίνεσα ε, Γιαλασέντερ ε, παλαιότερα ε, δεν έχουν έρθει σε επαφή με το Συμβούλιο. Δεν είναι το θέμα αυτό η έλλειψη επαφή. Το θέμα είναι ότι είμαστε σε ένα διαθεσμικό ε, καυγά σε εισαγωγικά. Οι απόψει είναι διαφορετικέ. Και βεβαίω όλα αυτά έχουν επιπτώσει και σε άλλα άλυτα θέματα που απτώνται και άλλων θεσμικών οργάνων. Νομίζω λοιπόν ότι για τούτη, το, για την έκθεση για την απαλλαγή θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε τη δική μας θέση ε, και βεβαίως έχουμε κάνει εμείς τη δική μας, ε, το δικό μας μερίδιο δουλειάς για την διαφάνεια οπότε ελπίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μία λύση μεταξύ μας. Αν δεν τα καταφέρουμε θα πρέπει να πάρουμε την νομική οδό. Η συγγήτρια τώρα είναι σημαντικός ο ρόλος της και βεβαίω θα υποβάλουμε και τις ε, τροπολογίες μας στην έκθεση. Να δώσουμε κλείνοντα λοιπόν το λόγο στην κυρία Τσέσκοβα και πάλι. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είπατε βασικά διάφορα πράγματα που συμφωνούμε την άποψή μου. Ίσως τα είπατε με διαφορετικά λόγια, αλλά τα ίδια πιστεύω. Με τα χαράς Άκουσα από τους συναδέλφους, σχεδόν όλους τους συναδέλφους, ότι υποστηρίζουν, ότι εγκρίνουν τη θέση μου. Υπάρχουν και τεχνικές νομικές λεπτομέρειες. Θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε ειδική ακρόαση γι' αυτό. Να συζητήσουμε το πώς υποτίθεται ότι θα πρέπει να χορηγούμε τις απαλλαγές προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τι πληροφορίες θα πρέπει να πετούμε, να ζητούμε, να μας χορηγούνται. Αυτό καταδεικνύει ότι η Επιτροπή μας έχει δικαίωμα να θέτει ερωτήματα και να λαμβάνει απαντήσεις. Διότι διαφορετικά όπως και άλλα θεσμικά όργανα που αντλούν χρήματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Αυτά είναι πληροφορίες που πρέπει να χορηγούνται στο κοινό, στον κόσμο. Όλοι υποστηρίξατε το ότι πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια. Ο Ζαν έθεσε κάποιο ερώτημα νομίζω. Γιατί Γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εν συγκρίση με το Συμβούλιο Κοιτάξτε, κατά παρελθόν μου ζητήθηκε να συντάξω δύο εκθέσει. Μία αφορούσε την απαλλαγή προ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η άλλη έκθεση αφορούσε απαλλαγή προ το Συμβούλιο. Βασιζόμενη επί της δηλώσεως της ε, νομικής υπηρεσίας είπαμε ότι το 2011 ότι η απαλλαγή το 2011 απαιτούσε τη σύνταξη μίας μόνο εκθέσεως. Διότι τα αποτελέσματα εμπεριέχονται όλα σε ένα δημοσιονομικό κεφάλαιο. Βάσει λοιπόν της συστάσεως αυτής, συνέταξα μόνο μία έκθεση. Εσυγκρίση με την αρχική πρόθεση να συντάξω δύο εκθέσεις. Και γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα δύο αλληλένδετα θέματα που περιέχονται σε αυτή την έκθεση. Από το 2012 και μετά, κάποιος άλλος, όχι εγώ, θα συντάσσονται δύο εκθέσεις. Μία έκθεση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μία έκθεση για το Συμβούλιο. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που εξαρτάται και από περαιτέρω αποφάσεις. στα πλαίσια του νέου δημοσιονομικού κανονισμού που θα εμπεριέχει δικούς του κανόνες. Τώρα έτσι έχουν τα πράγματα. Μία έκθεση που καλύπτει και τα δύο θεσμικά όργανα, τους δύο θεσμούς. Ευχαριστώ για τις απόψεις σας, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Είμαι απλώς μια ταπεινή συγγήτρια, αλλά είμαστε εμείς εδώ όλοι μαζί σαν επιτροπή. Και ο Πρόεδρος ακούει αυτά που λέμε και εκτιμώ πάρα πολύ τη στάση του, την τοποθέτησή του, διότι βάσει όλων αυτών θα μπορέσουμε να συζητήσουμε πραγματικά τη δική μας θέση στις διαδικασίες αυτές. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ενωμένοι γίνεται. Αύριο, όπως σας είπα, θα συναντηθώ με εκπρόσωπο της Ιρλανδικής Προεδρίας και ο πρόεδρος ε, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Σίγουρα δεν θα είναι κάτι εντελώς ανεπίσημο, θα σας ενημερώσω δεόντως για όλα όσα θα πούμε. Όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, όπως ξέρετε αυτό δεν είναι δική μου έκθεση, είναι έκθεση του συναδέλφου μου, ε, είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσω Στην έκθεσή μου εμπεριέχονται κάποια στοιχεία που αφορούν την υπηρεσία εξωτερικής δράσεως, αλλά μόνο σε σχέση με την χρήση πόρων που μεταφέρθηκαν από τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου προς αυτό, αυτή τη νέα υπηρεσία. Όσον αφορά τα 411 και τα 80 εκατομμύρια ευρώ, αυτά τα συγκεκριμένα ποσά τα εξέτασα μόνο σε αυτό το πλαίσιο. Στο πλαίσιο δηλαδή του προϋπολογισμού του Συμβουλίου και των πόρων που μεταφέρθηκαν από εκεί. Διότι πέρσι όταν συζητήσαμε την απαλλαγή για το Συμβούλιο, συζητήσαμε το διαχωρισμό των πόρων από τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου και των πόρων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από ό,τι θυμάμαι, το αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν κάπως ασαφές. Χαίρομαι λοιπόν που κουβεντιάζουμε το θέμα. Χαίρομαι που το συζητούμε. Κάποιος είπε ότι θα χρειαζόταν να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή, να εξεταστεί ξεχωριστά, πέρα από τη συζήτηση για τα άλλα θεσμικά όργανα. Άλλα θεσμικά όργανα όπως είναι η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ο Διαμεσολαβητής, το Ευρωπαϊκό Λεκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και άλλοι φορείς. Ευρωπαϊκός Επόπτης ε, Προστασίας των Δεδομένων, ξεχωριστά από όλα αυτά τα όργανα. Όλα αυτά υπόκειται στον έλεγχο της, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ακούστηκαν, ε, γράφτηκαν ελάχιστες επικρίσεις με την εξαίρεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και των διαδικασιών προσλήψεων που ακολουθεί. Όμως, λάβαμε απαντήσεις στις ερωτήσεις μας και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους όλων εκείνων των θεσμικών οργάνων που απάντησαν. Τους ευχαριστώ πραγματικά. Και ένας δύο συνάδελφοι αναφέρθηκαν επίσης και στον Ευρωπαϊκό Επόπτη των Προστασίας των Δεδομένων και στο διαμεσολαβητή. Κάποιος είπε ότι η διάρκεια των ελέγχων των ελεγκτικών διαδικασιών γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πολλοί λίγοι, ελάχιστοι Ευρωπαίοι πολίτες χρησιμοποιούν αυτόν τον φορέα το συνήγορο του πολίτη, τον διαμεσολαβητή. Και γι' αυτό πρότεινα κάποια μέτρα, μέτρα που αφορούν την προβολή αυτού του θεσμού. Έχω ένα άλλο σχόλιο που αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν εμπίπτει στη δική μου αρμοδιότητα, αλλά θα ήθελα κροθυγός να σχολιάσω. Θέλω να πω ότι από ό,τι φαίνεται έχει την παράδοσή του, έχει το βάρος του, μεγαλύτερες δαπάνες, αυτό είναι κάτι που δεν πειράζει, το μεγαλύτερο κόστος, όμως ελπίζω και εύχομαι όλα αυτά να αντικατοπτριστούν με κάποιο τρόπο σε γραπτές τροπολογίες που σίγουρα θα με βοηθήσουν. Έχω προφανώς λάβει γραπτές απαντήσεις. Κάποια, κάποιες φορές καταφθάνουν καθυστερημένα και εγώ ίδια θα έχω κάποιες τροπολογίες και ελπίζω και υποθέτω ότι ο κ. Τσαρνιέτσκι θα ακολουθήσει παρόμοιο μονοπάτι, παρόμοια προσέγγιση και ότι θα του προωθηθούν όλα αυτά τα σχόλια, θα τα διαβιβάσω και τα σχόλια και τις προτάσεις. Ελπίζω να έχω καλύψει τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και χαίρομαι που με αφήσατε να εκπροσωπήσω και το συνάδελφό μου που απουσιάζει για μία ακόμη φορά. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε καλές αποφάσεις. Προσβλέπω σε προτάσεις σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και για το χρόνο που μου διαθέσατε. Εγώ ευχαριστώ κύριε Τσέσκοβα. Κλείνουμε λοιπόν το σημείο αυτό και πάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Η απαλλαγή των οργανισμών. Πάμε στον κύριο Γκερμπράντι. Να του δώσουμε το λόγο κατευθείαν. Yes, thank you very much, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μέχρι τις 7.30 δεν έχουμε χρόνο, Πρόεδρε. Ωραία. Θα δούμε λοιπόν μέχρι πού θα φτάσουμε με 30 υπηρεσίες. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, για να θυμηθούμε λιγάκι το περί πρόκειται. Μιλούμε για, τις, ε, για τους οργανισμούς που ε, κάθε χρόνο πρικοδοτούνται με 1,3 δις. 750 εκατομμύρια εξ αυτών είναι δημόσια κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των οργανισμών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 10 χρόνια. Ξεκινήσαμε με περίπου 3 πριν από 10 χρόνια και τώρα έχουμε πάνω από 30. Οπότε είναι αρκετά σημαντικός ο αριθμός των οργανισμών. Πριν ξεκινήσω να σας αναφέρω και τις επιμέρους εκθέσεις αλλά και τις γενικές, ευχαριστήσω καταρχάς τους οργανισμούς για τη συνεργασία τους. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμη η βοήθειά τους. Πρέπει επίσης εδώ να πω ότι ε, δεν έχει υπάρξει τεράστια παρατυπία σε κάποιον από αυτούς τους οργανισμούς, οπότε Γενικώ πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί μας λειτουργούν. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια ειδικά επιμέρου σημεία για κάποιου επιμέρους οργανισμούς και υπάρχουν ε, και κάποια σημεία που θέλω να τονίσω από τις ε, οριζόντιες εκθέσεις που έχω κάνει. Ξεκινώντας. Πρέπει να τονίσω την ε, σημασία της ανεξαρτησίας αυτών των οργανισμών δημιουργήθηκαν από δουλειά βεβαίως που είχε γίνει ήδη από την Κομισιόν και για να, για να κάνουν αυτή τη δουλειά με πιο ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο. Υπάρχουν λόγοι ανησυχίας α, σχετικά με το ότι αυτή η, α, η ανεξαρτησία δεν είναι πάντα εγγυημένη και αυτό οφείλεται καταρχάς στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτούς τους οργανισμούς η Κομισιόν αλλά και σε πιο συστημικά προβλήματα. Για παράδειγμα, τα διοικητικά συμβούλια, όπου εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη. σε κάποιες περιπτώσεις ε, υπάρχουν, συγκρό... Ε, υπάρχουν συγκρόμενα συμφέροντα από τους εκπροσώπους των εθνικών ε, αντιπροσωπιών. Μιλούμε βεβαίω και για σύγκρουση συμφερόντων. Θα το κάνουμε και αργότερα μέσα στη βδομάδα, θα το συζητήσουμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και την σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του ίδιου του οργανισμού. Επίσης, άλλο ένα παράδειγμα, με, τα, με τις τρεις νέες υποπτικές, με τους τρεις νέους υποπτικούς οργανισμούς, όπου μία αξιολόγηση έδειξε ότι η ε, ανεξαρτησία τους θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερη από ό,τι είναι τώρα. Το δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω είναι η αποτελεσματικότητα των οργανισμών. Ξέρω ότι αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερο ευαίσθητο για τα κρατη αλλά ε, δεν είναι μόνο το ότι έχουμε πάει από τους 3 του 30 ε, οργανισμούς μέσα σε 10 χρόνια, αλλά έχουμε και αρκετούς οργανισμούς που είναι αρκετά μικρή σε μέγεθος. Και γι' αυτό πραγματικά αναμένω να συζητήσουμε ε, στην Επιτροπή μας τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ορίζει και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν ε, και στο μέλλον οι οργανισμοί αυτοί και επικεντρώνεται σε κάποια ίσως ενσωμάτωση επιμέρους οργανισμών σε έναν ή συγχώνευση κάποιων ή εν πάση ενίσχυση τη συνεργασία μεταξύ κάποιων οργανισμών. Υπό αυτό το φως λοιπόν θα ήθελα εδώ να σα προτείνω να προτείνουμε στους οργανισμούς αυτούς να, ε, διορίσουν έναν ε, ειδικό συντονιστή για τον ε, δικό χάρτη. Ξέρω ότι είναι, πολύ, είναι τεράστιο το καθήκον με πολλά σχέδια δράσης για όλους τους οργανισμούς. Ο οργανισμός που έχει αναλάβει την προεδρία ας πούμε, του δικτύου εξορισμού δεν είναι ανεξάρτητος, γιατί ουσιαστικά αποτελεί τμήμα του οργανισμού, αλλά θα, ίσως να, θα μπορούσαν ίσως να ε, διορίσουν έναν πρώην εκτελεστικό διευθυντή για να κάνει να αναλάβει το ρόλο του συντονιστή, ειδικά για τον οδικό χάρτη της Κομισιόν. Τρίτον, πάλι στα πλαίσια της οριζόντιας έκθεσης, το διοικητικό άχθος που έχουν να αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί. Σας έδωσα το παράδειγμα και κατά τη διάρκεια της ακρόασής μας, το Coffee Gate, όπως το, όπως το ονόμασα, είναι τεράστιο το, η χαρτούρα που έχει να αντιμετωπίσει ένας διευθυντής για να μου προσφέρει εμένα, ας πούμε, όταν τον επισκεφθώ, ένα, ένα, έναν καφέ. Το ίδιο ισχύει και για την απασχόληση, για τη διαδικασία διορισμών. Οι οργανισμοί δεν είναι σαν την Κομισιόν με δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Οπότε ίσως να πρέπει να αλλάξουμε τις διαδικασίες διορισμών τους, έτσι ώστε να ταιριάζουν καλύτερα αυτοί, αυτές οι διαδικασίες στη δουλειά που έχουν επιτελέσουν αυτοί οι οργανισμοί. Ένα τέταρτο σημείο στην έκθεσή μου είναι η σύγκρουση συμφερόντων την συζητήσαμε και κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Είναι σαφές ότι οι κατευθυντήρες γραμμές που χρησιμοποιούμε τώρα του ΩΣΑ δεν ταιριάζουν απολύτως στις ανάγκες των οργανισμών. Ας πούμε, οι, οι υπάλληλοι, μάλλον οι κατευθυντήρες του ΩΣΑ, μιλούν μόνο για υπαλλήλου. Πολλές ε, υπηρεσίες όμως χρησιμοποιούν ε, εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και αυτοί δεν καλύπτονται από τις κατευθυντήριες του ΩΣΑ. Και αυτό αναφέρεται και στον οδικό χάρτη της ε, Κομισιόν και όπως άκουσα και από την Κομισιόν θα πρέπει να έχουμε δικούς μας, δικές μας κατευθυντήρες γραμμές για να αποφύγουμε περιπτώσεις συγκρούσεως συμφερόντων στο μέλλον. Ένα τελευταίο σημείο που θέλω να τονίσω είναι η σχέση που έχουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτούς τους οργανισμούς. Έχουμε εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο, Έχουμε και αξιωματικού συνδέσμου. Α πούμε, εγώ είμαι ο συνδετικό κρίκο ε, για την Επιτροπή, για τον Οργανισμό για το Περιβάλλον. Αλλά και αυτό είναι πάλι σε μια ad hoc βάση. Βεβαίω πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη σχέση, καλύτερη επαφή με αυτού του οργανισμού, όχι μόνο για να αυξήσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία του, αλλά για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και την εμπειρογνωμοσύνη που, που έχουν αυτοί οι οργανισμοί εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, περνάω στις επιμέρους εκθέσεις. Όπως είπα στην αρχή, δεν υπάρχουν τεράστια προβλήματα που να βρέθησαν από το ελεκτικό συνέδριο. Βεβαίως υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία τονίζονται από το ελεκτικό συνέδριο. Ξεκινώντας, υπάρχει η γνωμοδότηση για το ECDC, για το ε, παρατηρητήριο ε, τοξικομανίας και ναρκωτικών ε, Υπάρχει η Συμφωνία Πλαίσιο, η οποία επίσης ε, ε, κοινοποιήθηκε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, με συγχωρείτε. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό είναι λόγος για να αναβάλουμε ή να απορρίψουμε την ε, απαλλαγή αυτού του οργανισμού. Επίσης, άλλη μία, άλλος ένας οργανισμός, στον οποίο θέλω να επικεντρωθούμε, είναι η ΣΕΠΟΛ, η Αστυνομική Ακαδημία. Έχει συζητηθεί αρκετά συχνά η Αστυνομική Ακαδημία. Έχουμε δει σημαντικά προβλήματα στο παρελθόν. Τα περισσότερα έχουν λυθεί από τον νέο κλειστικό διευθυντή. Αλλά προκύπτουν και νέα προβλήματα. Ένα εξ αυτών είναι το ότι πρέπει να αποχωρήσουν από, τα, από τις εγκαταστάσεις τους το Μάρτιο του 2014. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μετακομίσει η ΣΕΠΟΛ στη Χάγη και έτσι να συνδεθεί πολύ, πιο, πολύ περισσότερο με την Europol. τώρα, το αν θα συγχωνευτεί με την Europol ή όχι, μπορούμε να το συζητήσουμε. Ξέρω ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει συγκεκριμένη άποψη από αυτού. Αλλά τουλάχιστον υπάρχουν πάρα πολύ καλοί λόγοι, ειδικά σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα, για να μετακομίσει στην Χάγη η ΣΕΠΟΛ. Επίσης, άλλη μια, άλλος ένας οργανισμός είναι ο Οργανισμός των Μιλωδών Δικαιωμάτων. Έχουν υπάρξει κάποια προβλήματα τα τελευταία χρόνια που είναι περισσότερο προσωπικής φύσεως. Έχουμε δει κάποιους ε, εργαζόμενους να αντιμετωπίζουν προβλήματα με το Συμβούλιο, με τους διευθυντές τους, και θα ήθελα να δώσουμε τη δέωσα προσοχή σε αυτό γιατί φαίνεται να είναι κάτι παραπάνω από κάποιες απλές επιμέρους ή περιπτώσεις. Βεβαίως ε, ευχαρίστως να αναθεωρήσω την άποψή μου αν με πείσει κάποιος για το αντίθετο. Τώρα, τα θέματα ε, αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να υπάρξει στενότερη συνεργασία ως προς αυτά. Έχουμε τρεις ε, οργανισμούς που είναι αρκετά μικροί και ασχολούνται ακριβώς με το ίδιο θέμα, ακριβώς στον ίδιο τομέα. Οπότε νομίζω ότι θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε από μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ αυτών των τριών. Τέλος, Πρόεδρε, για, τις, για τους επιμέρους οργανισμούς έδωσα, προσοχή εγώ στις τρεις, στους τρεις οργανισμούς που για πρώτη φορά τους βλέπουμε στην ε, διαδικασία απαλλαγής, τους τρεις για το δημοσιονομικό έλεγχο. Μερικώς ε, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μερικώς από τα κράτη-μέλη. Στην επαφή που είχα με τους οργανισμούς και με το ελεκτικό συνέδριο, ε, φάνηκε ότι αυτή η διπλή μορφή χρηματοδότησης δεν είναι η πιο αποτελεσματική τελικά. Είδαμε κάποιες ε, έτσι, περίεργες περιπτώσεις με κάποια κρατημέλη. Είχαν ε, πρόβλημα στο να καταφέρουν να αποκτήσουν τα απαραίτητα κονδύλια. Ε, επίσης, να μην ξεχάσουμε τις κοινέ δράσεις που είναι κομμάτι αυτής της διαδικασία απαλλαγή. ο συνολικός προπολογισμό τους είναι υψηλότερο από, από, όλο το, από το σύνολο του προπολογισμού των οργανισμών. Για το, για το 2011 ήταν 877 εκατομμύρια. Ο συνολικός προπολογισμό για όλη τη διάρκεια ζωής τους είναι πολύ μεγαλύτερος ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει τεράστια εισρωή ιδιωτικών κονδυλίων ο συνολικός, η συνολική ε, επιδότηση της Ένωσης φτάνει τα 11 δις. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά το θέμα αυτό. Από το ελεκτικό συνέδριο είδαμε κάποιες ε, γνωμοδοτήσεις που κυρίως έχουν σχέση με συναλλαγές με μεμονωμένες επιχειρήσεις και είναι δύσκολο να εφαρμοστούν τα σωστά συστήματα έτσι ώστε να εγγυηθούμε την ε, καλή διαχείριση, την σωστή δαπάνη αυτών των κονδυλίων. Οπότε πρέπει να το δούμε αυτό. Άλλο ένα πρόβλημα είναι ο χαμηλός ε, ρυθμός πληρωμών είναι μάλιστα τόσο χαμηλά τα ποσοστά που πραγματικά πρέπει να ανησυχήσουμε για το αν αυτές οι κοινέ δράσεις ε, όντως εφαρμόζουν το πρόγραμμα που έχουν ε, αναλάβει μέχρι το 2017. Η μειωμένη χρήση του προπολογισμού είναι σοβαρό ε, πρόβλημα. Επίσης, ένα άλλο θέμα για το οποίο χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες είναι το ότι στην Ελλάδα υπάρχουν projects τα οποία θα πρέπει να λάβουν εθνική χρηματοδότηση, αλλά για κάποιο λόγο λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα διευθυντικά ταμεία. Και αναρωτιέμαι και θέτω το ερώτημα και στην Κομισιόν και στο Ελεκτικό Συνέδριο, γιατί συμβαίνει αυτό. Τέλος, Πρόεδρε, για να μην δαπανούμε άλλο χρόνο και για να μπορέσουν και οι συνάδελφοι να πούν την απόψή τους, δεδομένου του όγκου των κονδυλίων που δαπανώνται από αυτές τις κοινέ δράσεις και λόγω και της δομής που έχουν ως ε, συμπράξεις σε δημοσιοδητικού τομέα, ε, θα ήθελα να καλέσω το Ελεκτικό συνέδριο να κάνει μια ειδική έκθεση για αυτές ακριβώς τις κοινέ επιχειρήσεις και να δει την αποτελεσματική ή μη εκτέλεση των προγραμμάτων σχετικά και με την έρευνα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Γκερμπράντη. Ένας θέλει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε εισηγητά, για την ε, δουλειά που κάνατε για να εξοικονομήσω χρόνο. Καλό θα ήταν να συζητήσουμε βέβαια και λίγο και μπαίνω στο ψητό. Το εξή. Ποια είναι η ουσία, ο πυρήνας, ποιος είναι ο ρόλος, ποιες είναι οι ευθύνε του Κοινοβουλίου όταν χορηγεί απαλλαγή ή όταν δεν τη χορηγεί σε διάφορους οργανισμούς ανεξάρτητα από την απάντηση του καθενός, ρόλος είναι να προσέχει το Κοινοβούλιο με μεγάλη προσοχή το πώς διατίθεται τα χρήματα του φορολογουμένου. Σύγκρουση συμφερόντων και διαφάνεια είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Θα το έχετε ξανακούσει αλλά θέλω να σας δώσω κάνα δύο παραδείγματα. Γιατί θεωρώ ότι θα έχω πολλές τροπολογίες να υποβάλω και την οριζόντια έκθεση χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα και την, Ευρωπαϊ... την έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και την έκθεση της. Οριζόντια έκθεση πρώτα απ' όλα. Είναι το βασικό έγγραφο κατά κάποιο τρόπο. Άρθρο 19 λέει ότι εκφράζει τη λύπη της ...σύμφωνα σύμφωνα τα απορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου τη στιγμή ολοκλήρωση των επιτόπιων ερευνών για την σύνταξη της ειδική εκθέσεως Οκτώβριο του 2011 κανένας από τους τέσσερις επιλεχθέντες οργανισμούς κατάφερε να χειριστεί σωστά σύγκρουση φερόντων. Η MAA και η FSA είχαν αναπτύξει πιο προχωρημένες πολιτικές για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων κλπ. λοιπά. Εγώ τι έχω να πω. Αν είμαστε εμείς ικανοποιημένοι με τη σημείωση αυτή ότι η FSA έχει πια ανεπτυγμένες πολιτικές για τη διαχείριση του θέματος των συγκρούσεων συμφερόντων, αν εκεί αρκεστούμε, δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί, να σας πω γιατί. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας Τροφίμων. Σχέδιο εκθέσεως. Άρθρο 7 και άρθρο 9.2. Άρθρο 7. Λέει. Εκφράζεται η λύπη διότι σύμφωνα κλπ. κλπ. βασικά αυτά που προανέφερα. Σημειώνεται όμως ότι ο οργανισμός ανέπτυξε ήδη προχωρημένες πολιτικές για τη διαχείριση συγκρούσεως συμφερόντων. Συζητούμε συζητούμε κατά πόσο θα χορηγήσουμε απαλλαγή για το έτος 2011, για το οικονομικό έτος 2011, όταν ξέρουμε ότι είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει ε, τρόπος διευθετήσεως ε, συγκρούσεως συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας Τροφίμων. Τον περασμένο Αύγουστο είχαμε μία υπόθεση με το Διεθνές Ινστιτούτο Ζωντανών Επιστημών, ILSI, και ένα μέλος της ΕΦΣΑ, της δίκης της ΕΦΣΑ, ήταν μέλος και το ILSI. Όταν η ΕΦΣΑ ελέγχθηκε και ζήτηθηκε να απαντήσει, μας είπε «Έχουμε νέα πολιτική ανεξαρτησίας». Και αυτή η δραστηριότητα, δεν να είναι κανείς μέλος και του Διεθνούς Ινστιτούτου Ζωντανών Επιστημών της Επιστημονικής Επιτροπής εκεί και ταυτόχρονα να είναι μέλος με τον ίδιο ρόλο στο πάνελ της ΕΦΣΑ είναι κάτι συμβατό και ταιριάζει με τη νέα πολιτική ανεξαρτησία του οργανισμού. Τι σημαίνει αυτό? Ο φορολογούμενος θα ρωτούσε τότε ποιος κοιτάει κατά πόσο η πολιτική αυτή της ανεξαρτησίας έχει κάποιο νόημα και εγώ ρωτάω, αν δεν είμαστε εμείς, τότε ποιος είναι. Κανένας. Νοέμβριος 2012. Γενετικά τροποποιημένα έντομα και αξιολόγηση κινδύνου που δημιουργούν τα έντομα αυτά. Ομάδα εργασίας της EFSA συμπεριλάμβανε πολλούς εμπειρογνώμονες που είχαν άμεσες σχέσεις με την Oxitec. Η Oxitec είναι η εταιρεία η οποία αναπτύσσει αυτή τη μέθοδο. Τα γενετικά τροποποιημένα έντομα. Δεκέμβριος 2012. Le Monde αναφέρει ότι 8 από 18 μέλη της ομάδας εργασίας της CFSA για διάφορους συντελεστές που δημιουργούν προβλήματα ενδοκρινικά είχαν ε, θέσει τέτοια που οδηγού σύγκρουση συμφερόντων με αυτό το τομέα. Και όταν ρωτήσαμε την ΕΦΣΑ, η ΕΦΣΑ είπε δεν υπάρχει πρόβλημα. Και δεν άλλαξε τη σύνθεση της ομάδας εργασίας. Αυτά κάποια παραδείγματα, θα σας εξαντλήσω με άλλα παραδείγματα. Βέβαια υπάρχουν και άλλες εκθέσεις και δεν έχω προβλήματα με τις περισσότερες από αυτές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας Τροφίμων, η EFSA, δεν αγγίχτηκε σε αυτή τη συζήτηση μέχρι τώρα. Αλλά δείχνω αυτά τα παραδείγματα που παρέθεσα ότι πρέπει να συζητήσουμε ενδελεχέστερα το τι τρέχει εκεί, σε αυτόν τον οργανισμό. Άλλο παράδειγμα, το οποίο θέλω να παρουσιάσω και μετά θα το βουλώσω, είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Τι να πω, είναι παράξενο που στην έκθεση, στο σχέδιο εκθέσεως, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει όσον αφορά τη συνέχεια που έχει δοθεί στα όσα συζητήσαμε πέρσι. βάση για το όλο εγχείρημα είναι η συνέχεια που δόθηκε μετά την απαλλαγή του 2010. Γιατί δεν υπάρχει καν ίχνος συνεχιζομένων συνεχιζόμενα προβλήματα συγκρούσεων συμφερόντων και διαφανείας όσον αφορά αυτόν τον οργανισμό ένα εκατομμύριο ευρώ σύμβαση πλαίσιο με μια εταιρεία παραγωγής βίντεο που δεν υπάρχει πια. Πριν από κάποια χρόνια υπεγράφει σύμβαση και μετά ανανεωνόταν ετησίως και το 2011 που είμαστε τώρα και μιλάμε και συζητάμε αυτή η σύμβαση ανανεώθηκε και μιλάμε για 271.000 ευρώ και το πλαίσιο το γενικό είναι ένα εκατομμύριο και δεν υπάρχει εταιρεία. Και όταν ρωτήσαμε τον οργανισμό, Γενικός Διευθυντής, η Γενική Διευθύντρια πέρσι μας είπε στις υπηρεσίες περιβάλλοντος δεν έχουμε σύμβαση με την εταιρεία των βίντεο στην Κοπενχάγη, αυτή που συζητούμε. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα διότι η σύμβαση που υπεγράφει συνήθει με εταιρεία που δεν υφίσταται, που δεν έχει παράγει τίποτα, ούτε δευτερόλεπτο βίντεο δεν έχει παράγει και μιλάμε για ένα εκατομμύριο ευρώ. Και δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα στην έκθεση, καμία αναφορά. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο τώρα γι' αυτό, αλλά θα ήταν καλό να ακούσουμε κάτι. Κάποια λογική, κάποιο λόγο, κάποια τελόγηση. Τα coffee gates οι παρατηρήσεις για τα τύπου Coffee Gate που ακούστηκαν. Τα σχόλια τέτοιου τύπου που αποκαλύπτουν σκάνδαλα και προβλήματα είναι απαραίτητα, όπως και αυτά που λέω τώρα. Και θα πρέπει ισότιμα να τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Να εξετάζουμε με κριτικό όμα τις συγκρούσεις συμφερόντων και τα θέματα διαφανείας εφόσον προβληματιζόμαστε για άλλα θέματα. Πώς να μειώσουμε τα προβλήματα τα χρονικά, να μειώσουμε το χρόνο που ε, χρειάζονται από το χρόνο που χρειάζεται το ελεκτικό συνέδριο να ελέγξει αυτούς τους οργανισμούς. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε τι έγινε με τα περσινά προβλήματα, πώς εξελίχθηκαν. Να μην τα αφήσουμε πίσω, διότι ταυτόχρονα δεν εξυπηρετείται καν και το συμφέρον των οργανισμών αυτών, εάν αφήνουμε τα προβλήματα πίσω. Και σίγουρα δεν εξυπηρετείται το συμφέρον του φορολογουμένου. Όντας και εγώ φορολογούμενος, διερωτώ με Πώς μπορούμε να λησμονούμε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε πέρσι με αυτούς τους οργανισμούς. Δεν νομίζω ότι έχουν λυθεί ακόμα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Βαλτσίτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρου της συναδέλφου μου, τη κυρία Αγιάλα Σέντερ, που είναι σκιώδης εισηγήτρια για αυτά τα σημαντικά, πολύ σημαντικά έγγραφα και ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση και μου ζήτησε να εκφράσω την θέση της ομάδας S&D. Υποστηρίζουμε τα σχόλια που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα και, τις, και συγκεκριμένες τροπολογίες ε, θα υποβληθούν εντός των προθεσμιών. Και τώρα κάποια προσωπικά σχόλια που θα ήθελα να εκφράσω. Νομίζω ότι είναι ευπρόσδεκτο το ότι αυξήθηκε ο αριθμός των οργανισμών από 3 σε 30. Μπορούμε να εστιαστούμε επί των λειτουργιών αυτών των οργανισμών η γενική δομή έχει περιπλακή και πρέπει να αξιολογήσουμε το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα των φορολογουμένων. Όμως, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι οι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για κάποιους συγκεκριμένους προκαθορισμένους τομείς και τα αποτελέσματα ετησίως βελτιώνονται. Βλέπουμε από τις εκθέσεις ότι κάποιες ελλείψεις ε, έχουν καλυφθεί. Επίσης, υπάρχουν και πολύ σημαντικά ερωτήματα, σημαντικοί τομείς ε, που βελτιώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ισοτιμία των δύο φίλων, ε, η ισότητα των φύλων είναι πάρα πολύ σημαντική για όλα τα κράτη-μέλη. Είναι δύσκολη η διαδικασία που ακολουθείτε, προχωρούμε όμως. και αρκετά έγγραφα έχουν ε, αναφέρει το θέμα των συγχωνεύσεων του Ινστιτούτου και του Οργανισμού για την Ισότητα των Φύλων. Θα πρέπει αυτό το θέμα να το υπογραμμίσουμε και να αποφύγουμε την κατάσταση κατά την οποία και οι δύο φορείς θα παραλύσουν εν αναμονή της συγχωνεύσεως. Αυτά είναι τα σχόλια που έχω. Και συγκεκριμένες τροπολογίες θα, θα υποβληθούν αργότερα στον εισηγητή. Jean-Pierre. Ο jean όχι. Ωραία, αποσύρθηκε. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών εδώ. Να δώσω τον λόγο στον εισηγητή και πάλι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Κεμπατσίτης και τον Σέβαραν για τα σχόλιά τους. Ε, καλωσορίζω όλος ιδιαίτερος την κριτική στάση του κ. Σαφμαέρ. Ε, συμφωνώ απόλυτα με ε, το ποιος είναι ο βασικός μας ρόλος, η ουσία του ρόλου μας στη διαδικασία της απαλλαγή. Θα ήθελα να το θέσω και πιο στεναρά. Είναι η μόνη χρονική περίοδος που ελέγχονται οι οργανισμοί κάθε χρόνο. Μην υποτιμούμε λοιπόν το ρόλο που παίζουμε. Μιλάμε για 750 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Άρα παίρνω το ρόλο μας πολύ στα σοβαρά. Τα δύο σημεία που αναφέρατε πιο συγκεκριμένα, σύγκρουση συμφερόντων και διαφάνεια. Συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε εξετάσει επί σειρά ετών το πρόβλημα της σύγκρουσης συμφερόντων από το 2009 που ξεκίνησα την καριέρα μου στο Κοινοβούλιο όλο και κάποτε το συζητούσαμε, εγώ ζήτησα να γίνει βασική συζήτηση επί της συγκρούσεως συμφερόντων εντός των οργανισμών και όχι ad hoc. Αν υπήρχαν βασικές αποφάσεις από οργανισμούς όπως η ΕΦΣΑ, έβλεπες από διάφορες πλευρές του Κοινοβουλίου ε, να, από διάφορες ομάδες να θέτουν το πρόβλημα της συγκρούσεως συμφερόντων χωρίς να εξετάζει το πυρήνα του προβλήματος. Δηλαδή γενικά φιλοσοφικά το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Και είχαμε συζητήσει σοβαρά το θέμα, πολύ σοβαρά. Σύγκριση ΕΦΣΑ με τους διαφόρους οργανισμούς που κάνουν τη δουλειά στις ΗΠΑ. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργαζόμαστε με εξωτερική τεχνογνωσία η οποία προσλαμβάνεται. Και το να βρίσκουμε 100% ανεξαρτήτους με τις αναγκαίες ε, δεξιότητες να το κάνουν αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Κάποιες διασυνδέσεις υπάρχουν με πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή έρευνα. Ε, προσπαθήσαμε μέχρι τώρα, δεν το πετύχαμε 100%, συνεχίζονται οι προσπάθειες, θέλουμε να γίνουν διαδικασίες ε, όσο πιο ξεχωριστές, όσο πιο διαφανείς, όσο πιο ανεξάρτητες γίνεται, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε ε, συγκρούσεις συμφερόντων. Δεν φτάσαμε εκεί. Το 100% είναι αυταπάτη. Πρέπει να στεστούμε από αυτού. Ε, ήμουνα πολύ ικανοποιημένος με τις ε, απαντήσεις του Διευθυντού της ΕΦΣΑ στην ε, ακρόαση που αναφέρθηκε στο, στη δρομολόγηση ενός πιλωτικού προγράμματος σε διάφορους τομείς για την πρόσληψη τεχνογνωσίας από μέσα από τον οργανισμό αντί να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί εμπειρογνωμόνες. Βέβαια αυτό είναι πολύ πιο δαπανηρό από το να προσλάβει κανείς ε, εμπειρογνώμονες απ' έξω. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε και εδώ και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και σε άλλες επιτροπές. Είμαστε πρόθυμοι να πληρώσουμε δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, ούτω ώστε να έχουμε σοβαρή εγγύηση ότι υπάρχει 100% ανεξαρτησία σε οργανισμούς όπως είναι η ΕΦΣΑ. Και δεν μιλάμε μόνο για την ΕΦΣΑ, μιλάμε για διάφορους οργανισμούς. Είναι πολύ καλό θέμα προς συζήτηση. Με την επερχόμενη ακρόαση της Πέμπτης, με βάση την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και τη συνέχιση της συζητήσεως, διότι είμαστε στην αρχή της συζητήσεως, θα δοθεί συνέχεια, συμφωνώ απολύτως. Βλέποντας όμως τι έγινε το παρελθόν, 2011, που είναι το βασικό μας θέμα σε αυτή την απαλλαγή. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δίκαιο να αναβληθεί η ε, απαλλαγή μόνο και μόνο για αυτό το θέμα που συζητούμε επί σειρά ετών και συνεχίζεται η συζήτηση. Το άλλο σχόλιο σας για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, το ότι δεν παρακολούθησε του σύνεγγιστά όσα έγιναν μετά την περσινή έκθεση, είναι το, ο εξή λόγος. Εγώ και η ομάδα μου δεν συμφωνούσαμε με αυτά που είχαν συμπεριληφθεί στην περσινή έκθεση. Βασιστήκαμε στο δημοσιονομικό κανονισμό και δικός μας ρόλος δεν είναι να παίξουμε το ρόλο ενός εισαγγελέα, αλλά ανεξάρτητα και πολιτικά να εξετάζουμε κατά πόσο αυτοί οι οργανισμοί έχουν εφαρμόσει τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον έχουν εφαρμόσει σωστά και κατά πόσο έκαναν τη δουλειά τους με έναν πολιτικό σορθό τρόπο. Και πέρσι ήμουν απόλυτα πεπισμένος ότι η υπηρεσία περιβάλλοντος δεν ε, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα. Περισσότερα μικρά προβλήματα διαπιστώθηκαν, τα περισσότερα από αυτά επελήθησαν πέρσι. Έγινε εντατικότατη συζήτηση επ' αυτού, εκτενής εξηγήσεις δόθηκαν από τον οργανισμό και από το ελεκτικό συνέδριο για τα θέματα αυτά τα οποία διαπιστώθηκαν ε, πέρσι και στην Ολομέλεια δείξαμε ικανοποίηση για τις ε, απαντήσεις αυτές και δώσαμε την απαλλαγή στη Σύνοδο στην ψηφοφορία το Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Και γι' αυτό δεν παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή αυτά τα ζητήματα. Κάλυψα κάποια θέματα τα οποία μας αφορούν. Μέχρι τώρα κύριε Πρόεδρε, μια σκήνη 7,5 7.30 ακριβώς, θα ήθελα να σταματήσω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά που τηρήσατε το χρονοδιάγραμμα, το κονδύλι το χρονικό. Τέλεια. Να υπογραμμίσω μια ιδέα που αναφέρατε. Ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας και την αρχή της αναλογικότητας που εμπεριέχεται και στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στη δουλειά που κάνουμε θα πρέπει αυτή την αρχή να την τηρούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους σας. Πέρα συνεδριάσεως, τα ξαναλέμε αύριο στις 9. Καλό σας βράδυ. Στις 9 λοιπόν και εδώ κλείνουμε τη συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ, καλό βράδυ.